Good afternoon, everybody. Χαίρετε. Θα σας παρακαλούσα να καθίσετε. Good afternoon. I'd like to... Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω όλους στην ακρόαση. Αυτή για τη μείωση των εθνικών εκπομπών μετά το 2020. Πρέπει πρώτα να σας πω γιατί προεδρεύω ως εισηγήτρια. Δεν ήθιστε αυτό αλλά ο κύριος Λαβία, ο πρόεδρος ε, ε, κολλείεται. Ε, έπρεπε οπωσδήποτε να αποχωρήσει και ζητεί συγγνώμη γι' αυτό και ζητεί την επίοικιά σας. Ελπίζω να με ανεχθείτε ως πρόεδρο. Έτσι και αλλιώς εδώ θα καθόμουν, οπότε ανέλαβα και να προεδρεύσω. Σας καλωσορίσω όλους, ιδιαίτερα όσοι δεν είστε τακτικοί επισκέπτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. ευχαριστώ που ήρθατε, χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω εξ ονόματος ε, ε, της κυρίας Ντάλη που είναι μέλος και είναι εδώ μπροστά ε, να καλωσορίσω μια ομάδα φοιτητών από το Πανεπιστήμιο Λουφάν από τη Γερμανία. Καλωσορίσατε και ελπίζω να σας ενδιαφέρει η ακρόαση που θα ακούσετε συνέχεια. Λοιπόν, είναι μια κλασική ακρόαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ακούσουμε μερικές παρουσιάσεις και μετά ε, θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και απαντήσεις από τα μέλη και μετά θα ακούσουμε το δεύτερο πάνελ. Λοιπόν, προχωρώ αμέσως και δίνω το λόγο στο πρώτο πάνελ για θέματα υγείας και περιβαλλοντικά στην, στον έλεγχο της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. Για 10 λεπτά περίπου θα πάρει τώρα το λόγο η κυρία Μαρία Βεγού που θα μας μιλήσει για θέματα της ανθρώπινης υγείας για ε, τη βελτίωση της στο περιβάλλον της Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι αρμόδια στο Ευρωπαϊκό Κέντρο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας ε, για την ποιότητα, το αέρα και το θόρυβο. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και σας χαιρετώ όλους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και ηγείται η ΠΟΗ τα τελευταία χρόνια και παγκοσμίω, αλλά και στην περιφέρεια Ευρώπη. Ε, θα ήθελα σήμερα να σας παρουσιάσω αυτά τα τρία που βλέπετε στη διαφάνεια. Τι γνωρίζει η επιστημονική κοινότητα για το πώς επηρεάζει η ατμοσφαιρική ρήπανση την ανθρώπινη υγεία, πώς έχει κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να σας δώσω και κάποιες προοπτικές για τα ωφέλη ε, στην υγεία των Ευρωπαίων πολιτών αν μειωθεί η ατμοσφαιρική ρήπαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γιατί η μείωση εκπομπών ε, είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι ο υπαριθμόν ένα ε, υπέτειος παράγοντας για πρόορους θανάτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ε, άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους πρόωρα στην Ευρώπη λόγω της έκθεσης στην ατμοσφαιρική ρήπανση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Ο κόσμος αρρωσταίνει από την έκθεση στην ατμοσφαιρική ρήπανση στις πόλεις και σε πολλά μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα όχι μόνο αρρωσταίνει αλλά και πεθαίνει. Και υπάρχουν στοιχεία πάρα πολύ ε, εύγλωτα που λένε ότι η ατμοσφαιρική ρήπανση προκαλεί καρκίνο, αναπνευστικά νοσήματα και καρδιαγγειακά. Σας δείχνω εδώ αυτή τη γραφική παράσταση για να καταλάβετε με αυτή την εικόνα πώς οδηγεί ε, η ατμοσφαιρική ρήπανση σε σοβαρά προβλήματα υγείας. Όταν αναπνέουμε μολυσμένο αέρα, υποθέτουμε ενστικτοδός ότι επηρεάζει το αναπνευστικό και τους πνεύμονες, αλλά τα αιωρούμενα σωματίδια που είναι πάρα πολύ μικρά και αόρατα για το μάτι, μπαίνουν πολύ βαθιά στους πνεύμονες και καταλήγουν στην κυκλοφορία, στις αρτηρίες, στις φλέβες και μπορούν να περάσουν σε διάφορα όργανα του οργανισμού και να επηρεάσουν και το νευρικό σύστημα ε, και το αναπαραγωγικό, το γεννητικό σύστημα και το έμβριο ε, και ε, ακόμα σε έμβρια και σε νεογνά και πολύ μικρά παιδιά ε, νήπια μπορούμε να έχουμε προβλήματα και καρδιαγκιακά και αναπνευστικά. Δεν είναι λοιπόν ότι αναπνέω βρώμικο αέρα και έχω πρόβλημα στον πνεύμονα και στο αναπνευστικό μου. Είναι πολύ ευρύτερο. Εδώ ε, η επόμενη διαφάνεια σας δείχνει πώς η ατμοσφαιρική ρήπανση προκαλεί βλάβη στην υγεία και πόσοι πλήττονται. Συνήθως θεωρούμε ότι ο κόσμος πεθαίνει προώρα έτσι ονομάζεται και αυτό είναι ε, η κορυφή της πυραμίδας. Ε, αυτό μπορούν να το μετρήσουν καλύτερα οι κυβερνητικές αρχές ε, γιατί υπάρχει ένα μητρό που καταγράφονται με τις λεξιαρχικές πράξεις θανάτου και ξέρουμε πόσοι είναι νεκροί. Αλλά υπάρχουν πολύ περισσότεροι που επηρεάζονται και έχουν προβλήματα υγείας, δεν είναι μόνο οι θάνατοι. Κατεβαίνοντας λοιπόν αυτή την πυραμίδα ε, μπορεί να είναι οι βλάβες λιγότερο σοβαρές, ε, αλλά επηρεάζουν και πλήττουν περισσότερους ανθρώπους. Αυτό έχει να κάνει με την πνευμονική λειτουργία, καρδιακιακά, διάφορα αναπνευστικά σύνδρομα. Όλοι γνωρίζουμε κάποιον, ένα παιδί ή ένα συγγενή που έχει αναπνευστικά προβλήματα. Όταν έχει νέφος ή ε, θαλομύχλη. Αλλά υπάρχουν και άλλα πολλά ζητήματα υγείας, δεν είναι μόνο τα αναπνευστικά. Στον αστικό πληθυσμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο κόσμος εκτίθεται σε υψηλά επίπεδα βλαβερές συνέπειες και εδώ βλέπουμε διαφορά ανάμεσα στις οριακές τιμές και ε, τις κατευθυντήριες γραμμές της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Βλέπετε λοιπόν διάφορες χημικές ουσίες αριστερά και αιωρούμενα σωματίδια που ε, ρηπαίνουν τον ε, αέρα. PM2,5 που είναι πάρα πολύ ψηλά ε, σωματίδια που μπαίνουν μέσα στους πνεύμονες. Κοιτάξτε τα στάνταρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 10 με 14% του πληθυσμού ε, που εκτίθεται σε επίπεδα περισσότερο. Ενώ αν δείτε τις κατευθυντήριε γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αυτό φτάνει στο 91-93% του πληθυσμού που εκτίθεται σε βλαβερά επίπεδα. Είναι ευρύτερο το πρόβλημα, ευρύτατο. Δεν είναι μόνο κάτι που συμβαίνει στην Ασία ή στην Κίνα ή που τα βλέπουμε στις ειδήσει για άλλε χώρες. Ισχύουν και συμβαίνουν εδώ, στην Ευρώπη. Ε, αυτός ο χάρτης ε, είναι από μία έκθεση που δημοσιεύτηκε ε, πολύ πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Ε, νομίζω ότι θα το βρείτε εδώ στην αίθουσα, στην είσοδο, πώς έχουν τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε σκούρο πράσινο μερικές κουκίδες που είναι τα μόνα μέρη που ανταποκρινόμαστε στις συστάσεις του ΠΟΕ ως προς την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Θα πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα. Αν έχω να σας δώσω ένα μήνυμα, είναι ότι και μπορεί να βελτιωθεί η ατμοσφαιρική ρήπανση. Οποιαδήποτε βελτίωση του ατμοσφαιρικού αέρα θα οδηγήσει και σε βελτίωση της υγείας μας. Αυτό είναι πάρα πολύ ισχυρό επιχείρημα. Δηλαδή οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται, που θα έχουν αντίκτυπο και θα μειώσουν την ατμοσφαιρική ρήπανση, ε, αμέσως βελτιώνουν την υγεία. Ποιε είναι οι προοπτικέ για την Ευρωπαϊκή Ένωση για βελτίωση. Γνωρίζετε όλο το πακέτο για τον καθαρό αέρα και τα διάφορα αποτελέσματα που προτείνονται εάν εφαρμοστεί σωστά θα προλάβουμε πολλούς θανάτους και θα αποτραπούν μέχρι το 2030, θα μειωθεί ε, η στατιστική μείωση του προσδόκιμου ζωής. Δηλαδή περίπου 9 μήνες ε, λιγότερο ζουν σήμερα οι άνθρωποι λόγω της ατμοσφαιρικής ρήπανσης και αυτό θα μειωθεί στους 5,5 περίπου. Αυτό βελτίωση είναι και θα βελτιωθεί η υγεία του πληθυσμού. Θα είναι δωδεκαπλάσιο το κέρδος από το κόστος που θα έχουμε για τον περιορισμό. Δηλαδή συμφέρει και όλες η επένδυση αν θέλουμε να βελτιώσουμε τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Και μιλάμε για κόστος της τάξης από 40 μέχρι 140 δισεκατομμύρια σε εξωτερικό κόστος, αλλά ε, θα αυξαθεί η παραγωγικότητα του εργαζόμενου πληθυσμού, θα υπάρχουν λιγότερες ασθένειες και μάλιστα θα αυξηθούν και ε, οι θέσεις εργασίας, γιατί θα υπάρξει μεγαλύτερη παραγωγικότητα και ε, ανταγωνιστικότητα. Και αυτό είναι περίπου 0,02% του ΕΠ. Αρκεί αυτό άραγε. Όπως σας είπα προηγουμένως, οποιαδήποτε μείωση της ρήπανσης βοηθάει και ε, βελτιώνει την υγεία, άρα είναι θετική από μόνη της. Γνωρίζουμε όμως ότι υπάρχουν και άλλα τεχνικά μέτρα που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν ήδη από τώρα και ε, οι ε, Ευρωπαίοι αν τα υιοθετούσαν θα ζούσαν περισσότερο και καλύτερα. Τα όσα συζητούμε τώρα ε, στο 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον απέχουν πόρο από τις συστάσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για την υγεία γενικότερα, την ανθρώπινη υγεία και του περιβάλλοντος. Και επίσης απέχουν πολύ από τις κατευθυντήριες γραμμές για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Πολλά μπορούν να γίνουν για να βελτιωθεί η υγεία του πληθυσμού. Λοιπόν, θέλω να σας δώσω δεξής μηνύματα είναι σημαντικός παράγων ε, κινδύνου για τη ζωή μας, για την υγεία μας, παντού στον κόσμο και στην Ευρώπη η ατμοσφαιρική ρήπανση. Ε, ε, προκαλεί πολύ σημαντικές ασθένειες που έχουν μεγάλο επιπολασμό στον πληθυσμό, κάρδια, αναπνευστικά και καρκίνο του πνεύμονα. Η επιστημονική Κάνα στοιχεία ε, σωρεύονται και γνωρίζουμε για τον, τρόπο με τον οποίο επηρεάζει την υγεία η ατμοσφαιρική ρήπανση και πόσες ζωές χάνονται ε, εξαιτία αυτού και πόσους μήνες χάνουμε από τη ζωή μας λόγω της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Η έκθεση του ευρωπαϊκού πληθυσμού στη ρήπανση θα πρέπει να μειωθεί έτσι ώστε να βελτιωθεί η δημόσια υγεία. Είναι σημαντικό να επαναλάβουμε ότι οποιαδήποτε μείωση στην έκθεση θα έχει ευεργετικέ επιδράσεις στην υγεία. Η μείωση των εκπομπών από τι διάφορε πηγές είναι πολύ σημαντική και υπάρχουν ήδη σήμερα τεχνικά μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν. Γι' αυτό ελπίζω ότι θα γίνουν πολλά περισσότερα για να βελτιωθεί η ζωή όλων μας. Πραγματικά πιστέψτε με αυτά και σταματώ εδώ. ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε αμέσως στην περιβαλλοντική προοπτική και τις προοπτικές της ε, ποιότητας του αέρα στην Ευρώπη. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τώρα τον Κριστ Άγκρεν, που είναι διευθυντής ε, για την, υπεύθυνος για την ποιότητα του αέρα στο Airclean, στο Γκέτεμπορκ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Η οργάνωσή μου είναι ενεργό μέλος και στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος που έκλεισε τα 40 χρόνια, τα γιορτάσαμε πρόσφατα εδώ στις Βρυξέλλες, γι' αυτό είμαι εδώ στις Βρυξέλλες άλλωστε. Βλέπετε μια φωτογραφία εδώ, μια εικόνα μάλλον, του ενός κυνηγιού. Κυνηγάμε να πετύχουμε τους στόχους για το 2020 για να επαναλάβω αυτά που ακούστηκαν λίγο νωρίτερα. Υπάρχουν κάποιοι μακροπρόθεσμοι στόχοι και ο στόχος είναι να μην υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις και κίνδυνοι στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Αυτό είναι ο στόχος του προγράμματος περιβαλλοντικής δράσης και αυτό, αυτός ο στόχος τέθηκε και στο 7ο και στο 6ο πρόγραμμα και στο 5ο από τη δεκαετία του 90 χρονολογούνται αυτά. Οπότε ε, μπορούμε να επιστρέψουμε και να δούμε λίγο τα επιστημονικά δεδομένα όσον αφορά την προστασία με βάση την ε, καθοδήγηση του ΠΟΗ για την ε, προστασία των, οικοσυστημάτων, για την υπέρβαση των κρίσιμων επιπέδων και φορτίων για τα οικοσυστήματα και τη βιοπικιλότητα. Αυτές είναι οι συγκεντρώσεις, οι αναποθέσεις που πρέπει, στις οποίες πρέπει να επικεντρωθούμε για να βγάλουμε τα συμπεράσματα για το περιβάλλον. Τους έχουμε φτάσει αυτούς τους στόχους? Όχι. Αλλά βρισκόμαστε στον δρόμο προς τα εκεί. Εδώ βλέπετε την, ε, τις εκπομπές ε, διαφόρων ε, ατμοσφαιρικών ρήπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1990 έως το 2012. Κάποιες εκπομπές έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία 30 χρόνια. Από τη δεκαετία του 80 υπάρχουν ουσίες, συγκεκριμένα τα, τα οξύδια του θείου που έχουν μειωθεί κατά 90%. Τα οξύδια του αζότου κατά 50-60% η αμμονία μόνο κατά το 1 τρίτο και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην μεταρρύθμιση της ε, κοινή αγροτικής πολιτικής μετά το 1989. Δεν υπάρχουν όμως ε, τόσο σημαντικές μειώσεις όσον αφορά την αμμονία. Μια γρήγορη επισκόπηση να σας δώσω. Η υγεία είναι και αυτή ένα μέρος του περιβάλλοντος, οπότε θα σας επαναλάβω κάποια στοιχεία για την υγεία. Ε, μπορούμε όμως να δούμε εδώ και την οξύνηση, τους ε, ρήπους, ε, τους αζωτούχους ε, και τους θιούχους που μολύνουν το, το περιβάλλον. Υπάρχει επέρβαση των κρίσιμων φορτίων πάνω από 100.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα πλήττονται αυτή τη στιγμή των ε, ευαίσθητων οικοσυστημάτων. Επίσης, ε, η ζημιά που έχει κάνει η ε, ξύνηση τα τελευταία 40-50 χρόνια εξακολουθεί να υπάρχει. Θα χρειαστούν πολλές δεκαετίες ώστε να επανέλθουν τα οικοσυστήματα στην πρώτερη κατάστασή τους. Και περνάμε στον ευτροφισμό που είναι η υπερβολική χρήση λιπαν, λιπασμάτων από βιομηχανικές ε, ε, μονάδες στα ε, υδατικά και τα θαλάσσια συστήματα. Έχουμε ένα εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιόμετρα χερσαίων οικοσυστημάτων, περίπου το δύο, τα δύο τρίτα του Natura 2000 που έχουν μολυνθεί από αζωτούχες ενώσεις. Το 73% των περιοχών Natura 2000 πλήττονται. Επίσης υπάρχει το πρόβλημα του όζοντος που πλήττει ευαίσθητα φυτά και τα δάση, τις καλλιεργίες μας και τα υλικά, τα κατασκευαστικά. Και κάποιοι από αυτούς τους ρήπους έχουν αρνητικές επιπτώσεις και στην, στην πολιτιστική μας κληρονομιά που δεν τη συζητούμε πολύ ε, η αλήθεια είναι και δεν έχουμε ποσοτικά στοιχεία πολύ ε, εκτεταμένα. Αξίζει πάντως η επένδυση για την μείωση των ε, εκπομπών. Εδώ βλέπετε το, την υπερφόρτωση του, των οικοσυστημάτων. Εδώ μιλάμε για ολόκληρη την Ευρώπη σε αυτή τη διαφάνεια, ε, όχι μόνο για τις 28 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ε, εκπομπές ε, θείου είχαν, έφτασαν στο ανώτατο όριό τους ε, το 1990 και έχουν έκτοτε σημειωθεί σημαντικές μειώσεις της τάξης του 90%. Ε, παρόμοια στοιχεία υπάρχουν και για, την, ε, και τον ευτροφισμό και για την ε, οξύνηση. Τα οξύδια του, του αζότου και η αμμονία έχουν μειωθεί από το 1990 και εδώ μπορείτε επίσης να δείτε μια βελτίωση της απόθεσης δεν, δεν υπάρχει πλέον υπέρβαση των κρίσιμων φορτίων. Οπότε όταν μειώνουμε τις ε, εκπομπές η, το περιβάλλον ανταποκρίνεται όπως και η υγεία μας. Όταν σταματούμε να την εκθέτουμε σε αρνητικούς παράγοντες. Εδώ βλέπετε τη γεωγραφική κατανομή του ευτροφισμού και της οξύνησης τις περιοχές που πλήττονται από υπερβολικές ποσότητες αζωτούχων ενώσεων και θιούχων ενώσεων κάτω βλέπετε την, ε, ε, βελτίωση που θα ε, επιτευχθεί αν ε, επιτευχθούν στόχοι που έχουν ήδη τεθεί στο 2030. Έχουμε πολύ δρόμο όμως ακόμα μπροστά μας. Για την υγεία υπάρχει ένα παρόμοιο σενάριο, η τρέχουσα κατάσταση στα αριστερά, 2030 στα δεξιά και η προβολή για το 2030 το Βλέπετε εδώ την ε, μόλυνση από ατμοσφαιρικά σωματίδια 2,5 στις πιο σκοτεινές περιοχές του χάρτη. Εδώ είναι λίγο πιο σύνθετα τα πράγματα αλλά ε, η διαφάνεια αυτή δείχνει τα ίδια πράγματα. Ότι πάνω από 90% του αστικού πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτίθεται σε ε, επίπεδα όζοντος και ατμοσφαιρικών σωματιδίων που προκαλούν βλάβη στην υγεία. Δεν θα έπρεπε να μπορούμε να λύσουμε αυτά τα θέματα ε, ο καθένας μόνος του σε ένα βαθμό ίσως να γινόταν και αυτό. Κάθε περιοχή βεβαίως πρέπει να πάρει τα μέτρα της, αλλά αυτό δεν αρκεί. Πρόσφατα μια μελέτη ε, από, την, από τις Συμβούλες Κομισιών έδειξαν τις επιπτώσεις των διαφόρων πηγών ε, εκπομπής ε, σωματιδίων στις αστικές περιοχές σε κάθε κράτος μέλος. Εγώ πήρα ως παράδειγμα τις κάτω χώρες. Δεν είναι, το, δεν είναι το, το μέσο παράδειγμα, είναι ένα από τα ακραία παραδείγματα. Αλλά βλέπετε στην δεύτερη γραμμή, εκεί που λέει international, διεθνής, αυτό είναι η συγκέντρωση των σωματιδίων κατά μέσο όρο στις αστικές περιοχές στην Ολλανδία που εισάγονται από χώρες εκτός των, ε, της Ολλανδίας. Πάνω από το μισό της συγκέντρωσης σωματιδίων προέρχονται από ε, περιοχές εκτός της Ολλανδίας. Άρα η Ολλανδία δεν μπορεί με τίποτα να λύσει το πρόβλημα της μόνη της, το πρόβλημα το συγκεκριμένο. Πρέπει να υπάρξει συντονισμένη διεθνής ε, δράση. Και πολλές ε, πόλεις στην Ευρώπη συμβάλλουν στην ε, εκπομπή σωματιδίων και όζοντος και έχουν τέτοι, αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Οπότε πρέπει να συνδυαστούν οι διεθνή και τοπικά μέτρα για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Εδώ βλέπετε μια σχηματική αποτύπωση της, ε, των προτάσεων που έχουμε στο 2030. Βλέπετε το σενάριο αναφοράς. Εκεί ε, θα είμαστε αν εφαρμόσουμε την ισχύουσα νομοθεσία. Η πρόταση της Κομισιόν μειώνει τις εκπομπές, άρα μειώνονται και κατά λίγο οι επιπτώσεις. Δεν ε, όμως, δεν προβλέπει όμως η πρόταση Κομισιόν να την υλοποίηση όλων των τεχνικά εφικτών μέτρων για την επίτευξη των στόχων. Αλλά ήθελα να σας το δείξω αυτό. Θα ήθελα να, να σηκωθώ και να σας το δείξω και στον, και στον πίνακα. Αυτές οι προβλέψεις έγιναν πρωτού η, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει νέους στόχους για την πολιτική για το κλίμα. Φέτος τον Οκτώβριο η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να μειώσει το διοξείδιο του άνθρακα κατά 40% και να αυξήσει την ενεργειακή αποδοτικότητα και την συμμετοχή των ε, ανανεώσιμων. Με αυτόν τον τρόπο, αν ολιοποιηθούν, δηλαδή αυτά τα μέτρα, αυτόματα μειώνονται και οι εκπομπές ε, αζωτούχων και θιούχων ενώσεων και σωματιδίων. Και με αυτόν τον τρόπο το βασικό σενάριο που βλέπετε πάνω-πάνω πήγαινε πιο κάτω και την ε, γραμμή MTFR θα την κατέβαζε γιατί με τη μείωση αυτή θα, θα μπορούσαν να επιτευχθούν και, και νέα μέτρα. Τι έκανε λοιπόν η, η σύμβουλη, τι έκαναν οι σύμβουλοι της Κομισιόν σημαίνει ότι η πρόταση Κομισιόν τελικά είναι φθηνότερη από την εφαρμογή του σενάριου βάσης. Οπότε ε, εγώ συμπεραίνω ότι θα μπορούσαν να, να τεθούν ακόμη πιο φιλόδοξοι στόχοι με ακόμη μικρότερο κόστος από αυτό που αναμένεται. Αυτή είναι η πρόταση της Κομισιόν. Έχουμε δει μια σύνοψη. Ε, πρόκειται για τις μειώσεις ε, εκπομπών σε σχέση με τους παλιούς στόχους το κόστος είναι επιπλέον 3,3 δισεκατομμύρια κατ' ενώ το όφελος είναι τουλάχιστον δεκαπλάσιο. 3,3 δισεκατομμύρια κατ' όντως είναι πολλά χρήματα, αλλά αν το μοιράσετε στον ευρωπαϊκό πληθυσμό, μιλάμε για 6 ευρώ κατά άτομο κατ' Δεν είναι και τόσο δραματικά τα πράγματα δηλαδή και τα ωφέλη που ε, αποκομίζουμε είναι πολύ πολύ μεγαλύτερα. Εδώ βλέπετε τα περιβαλλοντικά αποτελέσματα της πρότασης Κομισιόν. Αν αν ακολουθούσαμε τους στόχους που είχε θέσει η Κομισιόν, θα, είχαμε, θα εξακολουθούσαμε να έχουμε 250.000 ε, πρόωρους θανάτους. Πάνω από τα μισά οικοσυστήματα ε, της Ευρώπης θα πλήττονταν από υπερέκθεση σε αζωτούχες και θειούχες ενώσεις και θα είχαμε προβλήματα υγείας που θα κόστιζαν ε, εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση και βλέπετε εδώ πόσο μακριά είμαστε ακόμα από τους μακροπρόθεσμους στόχους. Βλέπετε τι το CLE είναι οι τρέχοντες στόχοι, το NEC είναι η πρόταση της Κομισιόν και το MTFR είναι οι μέγιστες τεχνικά εφικτές τα μέγιστα τεχνικά εφικτά μέτρα. Και εδώ να σας πω τα συμπεράσματά μου. Νομίζω το βασικό συμπέρασμα είναι ότι τα προβλήματα στην υγεία και στο περιβάλλον είναι υπερβολικά μεγάλα και θα εξακολουθούν να είναι μεγάλα το 2030 και με την ισχύωση νομοθεσία και με βάση τις νέες προτάσεις της Κομισιόν. Νομίζω ότι η Κομισιόν και οι φορείς χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να θέσουν και να επιτύχουν τους στόχους που έχουν συμφωνηθεί ήδη πριν από 20 χρόνια. Και αν φτάσουμε εκεί δεν, θα, δεν χρειάζεται να έχουμε μόνο μια οδηγία για τα εθνικά όρια εκπομπών, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και νομοθεσία κατά κλάδο, ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα επιτευθούν μειώσεις εκπομπών στους σημαντικότερους τομείς και κλάδους. Στη γεωργία, Υπάρχει ένας τομέα μάλιστα που δεν καλύπτεται από την οδηγία αυτή που είναι οι διεθνέ μεταφορές όπου ε, οι εκπομπές αζωτούχων ε, αυξάνονται. Έχουμε την εγχώρια καύση στερεών καυσίμων που επίσης είναι μεγάλος παράγοντας μόλις και μια, και μια σειρά άλλων κλάδων. Και το σημαντικότερο είναι δεν αρκούν τα τεχνικά μέτρα. Χρειάζονται και πολιτικές. Οι πολιτικές για το κλίμα είναι πολύ σημαντικές και από τη σκοπιά της ε, ποιότητας του αέρα. Αλλά θα πρέπει επίσης να δούμε και τις πολιτικές για την ενέργεια και τις μεταφορές για να εξασφαλίσουμε ότι θα φτάσουμε στους στόχους μας έγκαιρα. Και εδώ στο τέλος να σας δώσω και μια ε, διαφήμιση, σας κάνω και μια διαφήμιση για το περιοδικό μας. Thank you. Thank you, σας ευχαριστώ που σεβαστήκατε το χρόνο σας. Περιμένουμε κάποιες ερωτήσεις από τα μέλη. Μάισνα. Πολύ γρήγορα μου δώσατε το λόγο. Α, στα αγγλικά. Δεν ξέρω αν έχετε στοιχεία για την ατμοσφαιρική ρήπαση ε, από ε, την αυσιπλοεία. Ε, δεν το βλέπουμε σήμερα. Εγώ είμαι από τη Βόρεια Ευρώπη και ξέρω ότι από την αρχή του 2015 ε, πρόκειται ε, για τη μείωση ε, την υποχρεωτική για τα σκάφη 0,01% θείου ας πούμε επιτρέπεται στη Βαλτική και στη Βόρεια Θάλασσα 0,05% στη Μεσόγειο. Έχετε στοιχεία για την ατμοσφαιρική ρήπαση από τα καυσαέρια των κουρασγερόπλιων, των ε, ποντοπόρων ε, πλοίων κτλ. Um, I can't Δεν μπορώ να σας δώσω αυτή τη στιγμή σε, ε, τονάζ της αποδόσεις, αλλά από το 1980 και μετά οι θιούχες εκπομπές αυξήθηκαν κατά ένα τρίτο και στο σύνολο των εμπορικών πλοίων κατά δύο τρίτα. Ε, ενώ όλες οι άλλες εκπομπές μειώνονται. Για τις θιούχες εκπομπές υπάρχει μια διαδικασία μείωσης η οποία θα φτάσει τα επόμενα χρόνια το 90% και από το 2020 θα υπάρξει επίσης και στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα και στην υπόλοιπη ε, βορειοανατολική θαλάσσια περιοχή αλλά δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ε, ιδιαίτερα αποτελεσματικά μέσα για τη μείωση των ε, οξυδίων ε, ζώτου και στις Ηνωμένε Πολιτείε υπάρχουν νέες ρυθμίσεις και τα νέα πλοία, οι νέες ναυπηγήσεις από το 2016 θα πρέπει να σημειώνουν μειώσεις εκπομπών οξυδίου αζότου 60% καλό θα ήταν αυτή η περιοχή ελέγχου να μην καλύπτει μόνο τις βόρειες περιοχές αλλά και τις ε, ε, νότιες και ε, βόρειο-ανατολικές επίσης. Να καλύψουμε έτσι συνολικά τις θαλάσσιες περιοχές γύρω από την Ευρώπη. Um, um, Σας ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη που έφτασα με καθυστέρηση. Ένα από τα θέματα τα οποία μου έχουν θέσει τα μέλη της κυβέρνησής μου είναι οι ανησυχίες που έχουν για τον έλεγχο, την παρακολούθηση και το τεράστιο κόστος το οποίο θα πρέπει να πληρώνουν οι διάφορες χώρες για τον σεβασμό της εφαρμογής των μέτρων αυτών. Θα πρέπει να γίνουν πολλά. Βλέπουμε ότι έχουν γίνει κάποια πρώτα βήματα στο σύνολο της Ευρώπης αλλά μπορείτε να μας πείτε πόσο συχνά κάνετε τις επιθεωρήσεις στον έλεγχο, ποιες υπηρεσίες παρακολουθούν και συλλέγουν τα στοιχεία. Γιατί αν είναι δυνατόν να γίνει μια σωστή μορφή παρακολούθηση τώρα, αυτό μπορεί να είναι ένα τεράστιο βάρος για ορισμένες χώρες. We already have Κοιτάξτε, υπάρχει έτσι και αλλιώ μια αντίστοιχη οδηγία κοινοτική για τα ανώτατα όρια η οποία εφαρμόζεται από το 2010, ψηφίστηκε για πρώτη φορά το 2001 έτσι ώστε οι εκπομπές ε, οι οποίες ελέγχονται, ε, αναφέρονται ε, και τα λοιπά. Ε, και στα πλαίσια του πρωτόκολλου του Κιώτου υπάρχει δηλαδή μια νομοθεσία καθρέφτης που δεν καλύπτει μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το σύνολο του κόσμου όπως και τη Βόρεια Αμερική. Ήδη από το 1999 υπήρξε αναθεώρηση το 2012 και υπάρχουν δεσμεύσεις για μειώσεις εκπομπών τουλάχιστον μέχρι το 2020. Έχουμε προσυπογράψει. Δεν έχει ακόμα επικυρωθεί ίσως, αλλά οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αποδεχθεί αυτές τις προτάσεις και δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε νέου τύπου μορφές παρακολούθησης και ελέγχου. Αυτό το οποίο ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να υπάρχουν κάπως πιο σύνθετα εθνικά προγράμματα έτσι ώστε οι μειώσεις των εκπομπών να γίνουν πραγματικότητα και να μπορέσουν να παρακολουθηθούν. Αλλά αυτό δεν είναι μια επιπλέον μορφή παρακολούθησης ή ελέγχου. Φυσικά αυτό συνδέεται και με την οδηγία για την ποιότητα του αέρα και αυτό έχει συμφωνηθεί από το 2008 και πρέπει να είναι εγκατεστημένη η μορφή ελέγχου ή έπρεπε τουλάχιστον να είναι από το 8. Οπότε επιπλέον κόστος, υπερβολικό κόστος δεν βλέπουμε που μπορεί να υπάρχει. Έχουμε μαζί μας κάποιον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω αν θα ήθελε να κάνει κάποιο σχόλιο. Είστε καλοδεχούμενος εφόσον το θέλετε αλλά δεν είστε υποχρεωμένος. Αν μπορείτε να βοηθήσετε στη συζήτηση αυτό θα ήταν χρήσιμο. Ευχαριστώ κύριε Γκέρλινγκ. Αυτό το οποίο είπατε είναι σωστό. Η νέα πρόταση δεν περιλαμβάνει νέες υποχρεώσεις ελέγχου είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως ευθυγραμμισμένο με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις και τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στα παλιά πρωτόκολλα. Ευχαριστώ Τζούντι. Ευχαριστώ και τους δύο μίλητες. Η ερώτησή μου είναι για ένα ειδικότερο θέμα είδα ότι υπήρξαν διαφορές στους στόχους ε, του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας ε, σε σχέση με τους αριθμούς τους οποίους προτείνουμε εμείς σαν Ευρώπη. Μπορείτε λίγο να μας εξηγήσετε πώς μπορούμε να μετακινηθούμε από εδώ που είμαστε σε εκεί που θα πρέπει να πάμε. Τα uh, Σχετικά με τα ιδιαιτέρως λεπτά σωματίδια, είναι ένας παράγον που μπορεί να έχει πάρα πολύ σημαντικές επιπτώσεις σε επίπεδο υγείας και αναρωτιέμαι πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Έχετε δίκιο οι διαφορές ανάμεσα στις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας για την ε, εκπομπή είναι 2,5, ε, είναι 10 μικρογραμμάρια, ενώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση το επίπεδο αναφοράς που θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ είναι 25 μικρογραμμάρια. Υπάρχει μια σημαντική διαφορά λοιπόν. Τα στοιχεία τα οποία έχει συλλέξει ε, ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας είναι θα έλεγα αρκετά πιστικά. Βλέπουμε εμείς πώς τα σωματίδια αυτά όταν αναπνέονται, όταν εισπνέονται μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα καρδιαγγειακά, αναπνευστικά κτλ. Τα παρακολουθήσαμε αυτά και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένε Πολιτείες. Και οι νέες μελέτες δεν περιορίζονται στα 10 μικρογραμμάρια αλλά πηγαίνουν και ακόμα πιο κάτω από αυτά. Λοιπόν, οι προτάσεις, ε, τα επίπεδα αναφοράς μάλλον του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας ε, βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία, ενώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν προηγηθεί πάρα πολλές συμβιβαστικές συζητήσεις, λαμβάνονται υπόψη στοιχεία όπως το εφικτό τεχνικά των μέτρων, οι ικανότητες των κρατών μελών να εφαρμόσουν τα μέτρα. Υπάρχουν δηλαδή και άλλα στοιχεία, άλλοι παράγοντες οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη όταν καθορίζονται τα επίπεδα αναφοράς που περιλαμβάνονται στις νομοθετικές ρυθμίσεις. Ενώ οι προτάσεις τις οποίες κάνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι προτάσεις. Σχετικά με τα υπερ σωματίδια, είναι πολύ πιο μικρά από τα PM25 στα οποία αναφερθήκαμε. Δεν υπάρχει σε επίπεδο Ευρώπης μια τέτοια μορφή παρακολούθησης. Είναι πάρα πολύ μακροπρόθεμο να παρακολουθηθούν σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Έχουν γίνει κάποιες μελέτες, έχουν βρεθεί κάποιες επιπτώσεις στην υγεία, αλλά βρισκόμαστε ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Πρέπει να υπάρξουν πολύ περισσότερες μελέτες έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε μέτρα τα οποία να μπορέσουν να εφαρμοστούν. Απαιτείται να γίνουν περισσότερα και η επιστημονική κοινότητα θεωρεί τα PM2,5 σαν τα σωματίδια, το ελάχιστο μέγεθος, τα οποία αφορούν κυρίως την υγεία. Αλλά θα πρέπει και με τα πολύ μικρού μεγέθου σωματίδια κάποια στιγμή να ασχοληθούμε επιστημονικά πρώτα. Ρωτήσατε και πώς μπορούμε να τα, να τα αντιμετωπίσουμε. Αυτό που γνωρίζουμε σήμερα είναι το εξής. Ε, ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστούν είναι να, υπάρχουν, να οριστούν κάποια όρια για τα οχήματα για να μην, ε, για, να, ε, και να διαθέτουν μια παγίδα για αυτά τα σωματίδια για τα, που πηγαίνουν στον αέρα στην ατμόσφαιρα από τα καυσαέρια. Ευχαριστώ κύριο Καπάντη. Ευχαριστώ, συγγνώμη που άργησα Απλά τώρα ε, κοίταξα λίγο τις διαφάνειες που παρουσιάσατε. Ελπίζω να μην ε, κάνω τώρα ερώτηση που έχετε ήδη ε, απαντήσει, πέραν των διαφανειών δηλαδή που παρουσιάσατε. Στη δημόσια συζήτηση μιλάμε συχνώς για τους πρόρους θανάτους, για το κόστος, το άμεσο και το έμεσο της ε, ατμοσφαιρικής ρήπανσης, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που εγώ το θεωρώ ίσως ακόμη πιο σημαντικό ή τουλάχιστον εξίσου σημαντικό. Και αυτό είναι οι επιπτώσεις που έχει η ατμοσφαιρική ρήπανση στην ποιότητα, του, την ποιότητα ζωής. Αν ένα παιδί δεν μπορεί να αθληθεί, για παράδειγμα, λόγω ε, του ότι πάσχει από ασθένειες που οφείλονται στην κακή ποιότητα ε, του αέρα. Αυτό έχει τεράστιες επιπτώσεις στη ζωή του και στην ποιότητα ζωής τους. Ίσως ε, έχετε κάποιες πληροφορίες και γι' αυτό το θέμα. Ε, θα μπορούσαμε τέτοιου είδους επιπτώσεις να τις ποσοτικοποιήσουμε με κάποιον τρόπο. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια. Ευχαριστώ. Έχετε δίκιο. Υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τους πρόωρου θανάτου, γιατί ακριβώς ε, είναι μετρήσιμο αυτό το στοιχείο. Υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία σε κάθε περιφάρεια, σε κάθε χώρα, οπότε μπορούμε να το μετρήσουμε, να μετρήσουμε συγκεκριμένα, τον αριθμό και είναι πάρα πολύ υψηλό, είναι δραματικά υψηλό. Αν και υπάρχουν πολλοί ε, διαφορετικές ε, ποικίλε ε, επιπτώσεις στην υγεία. Για παράδειγμα υπάρχουν άνθρωποι που πάσουν από άσθμα και σημαίνει παιδιά που δεν μπορούν να βγουν να παίξουν με τους φίλους τους. Και ε, υπάρχουν πληθυσμοί που πλήττονται από από την ζέστη και την ατμοσφαιρική ρήπανση ταυτόχρονα και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πολύ οξυμένα προβλήματα για κάποια τμήματα του πληθυσμού. Είναι πολύ πιο δύσκολο φυσικά να μετρήσουμε τα, αυτά που είπατε εσείς τις επιπτώσεις. Υπάρχουν κάποιες μελέτες και λεπτομερείς που έχουν ε, μετρήσει την επιπτώ, τις επιπτώσεις ε, της εθαλομίχλης ε, στην πνευμονική λειτουργία των παιδιών τις δύσκολες μέρες του καύσωνα για παράδειγμα, αλλά το να το παρακολουθούμε αυτό συστηματικά έχει αποδειχθεί ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και ο συνάδελφός μου εδώ ανέφερε στην παρουσίασή του ότι αυτό που συμβαίνει είναι ότι όταν ε, εξετάζουμε αυτά τα, τα στοιχεία πολλές φορές δεν βγαίνουν τα σωστά συμπερέσματα γιατί κοιτάμε μόνο τους θανάτους αλλά δεν κοιτάμε τις υπόλοιπες επιπτώσεις που βαρύνουν την, ε, που επιβαρύνουν την, την κοινωνία. Κοιτάμε την κορυφή του παγόβουνου, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που συνεπάρχουν, πάρα πολλές επιπτώσεις που συνεπάρχουν. mentioned... Σε μια φάση, συγγνώμη, η κυρία Ντάλη. Υπάρχει ένας κλάδος, είπατε, ε, των θαλάσσιων μεταφορών που αυτή τη στιγμή δεν διέπεται από κάποια νομοθεσία. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος ε, κλάδος που επίσης συνεισφέρει ε, όσον αφορά την κλιματική αλλαγή ε, και αυτός είναι, η αεροναυτιλία. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει νομοθεσία αλλά επαρκεί αυτή γιατί και αυτό το ερώτημα πολλές φορές ανακύπτει στη συζήτηση. Uh, έχω δει από τα στοιχεία. Οι αερομεταφορές δεν είναι ε, από τους μεγαλύτερους ε, υπετίους. Συνεισφέρει όντως, αλλά αυτά είναι πολύ ψηλά στον αέρα. Δεν είναι στην ατμόσφαιρα που εμείς αναπνέουμε. Και είναι πάνω από τα στρώματα εκείνα της ατμόσφαιρας που έχει ε, ανταλλαγές με το έδαφος, με τη γη. Είναι πολύ ψηλά. Όταν κάνετε μελέτη αντικτύπου για να διευρεθεί. Ε, να επεκταθεί ένα αεροδρόμιο. Το πρόβλημα και εκπομπέ δεν είναι τα αεροπλάνα, αλλά είναι τα αυτοκίνητα που πηγαίνουν έρχονται προς το αεροδρόμιο. Ε, αυτά για την αέρια κυκλοφορία και τα αεροσκάφη. Ε, ο αντίκτυπος εδώ είναι σε επίπεδο εδάφους, όχι τόσο ψηλά στην ατμόσφαιρα. Δύο σύντομε ερωτήσεις, η κυρία Μάισνερ. Είπατε ότι κυρίως Μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουν πολλές πόλεις. Λογικό είναι αυτό λόγω του αστικού πληθυσμού. Υπάρχουν πόλεις που είναι ε, ε, καλά παραδείγματα που έχουν βελτιώσει την κατάσταση. Οι κάτω χώρες είπατε ότι γενικά έχουν χειρότερο αέρα από άλλες περιοχές. Πώς γίνεται αυτό από τη θάλασσα, από τις γειτονικές χώρες, γιατί επειδή είναι κάτω από τη θάλασσα οι κάτω χώρες. Από περίεργεια ρωτάω. Μπορεί κάποιος Ολλανδός συνάδελφος να μου απαντήσει. Τώρα τι να απαντήσει κανείς, όλα ημικασίες μπορεί να κάνει κανείς. Είναι πολύ μεγάλη η πυκνότητα υψηλών εκπομπών στις κάτω χώρες και όχι μόνο και στο Βέλιο και στη Βόρεια Γαλλία ε, και στη Δυτική Γερμανία. Υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση ε, ε, ε, ρήπων και είναι και πολύ εντατική η θαλάσσια κυκλοφορία στα ανοιχτά. Δηλαδή και γύρω από την Ολλανδία και μέσα στη χώρα. Και επίσης από την εντατική γεωργία έχουμε εκπομπές αμμονίας που με ενώσεις και οξύδια και του θείου και του αζότου προκαλούν και παράγουν νητρικό αμμόνιο που είναι πάρα πολύ επιβαρυντικό. Είναι ένα συνδυασμός λοιπόν και τελικά καταλήγουμε σε υψηλές ε, συγκεντρώσεις αιρούμενων σωματιδίων στις κάτω χώρες. Γι' αυτό ο βασικός ε, λόγος είναι ε, η τόσο μεγάλη συγκέντρωση πορών ρήπων. Τώρα δεν έχω στο μυαλό μου καμιά πόλη που να έχει βελτιώσει σημαντικά την ατμοσφαιρική της ρήπαση. Τώρα Κάποιες οργανώσεις περιβαλλοντικές εκπονούν ένα οδηγό ε, City Ranking Guide, κάνουν μια κατάταξη δηλαδή των πόλεων σε ένα τέτοιο οδηγό και κοιτάνε ποιες πόλεις έχουν ε, ε, υιοθετήσει πολλά μέτρα. Υπάρχουν και βέλτιστες πρακτικές και καλά παραδείγματα σε πόλεις, αλλά έτσι δεν έχω τώρα στο μυαλό μου κάτι συγκεκριμένο. Να προσθέσω ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος έχει πολλά στοιχεία και έχετε στη διάθεσή σας μια έκθεση εδώ στην είσοδο ε, για εθνικά στοιχεία. Όχι βέβαια πόλη, αλλά χώρο σίγουρα μπορείτε να το κοιτάξετε. Και γεωγραφική κατανομή και ποια είναι η διαφορά από χώρα σε χώρα για τους ρήπους και ποιες οι τάσεις. Ευχαριστώ. Mm, Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω πολωνικά. Έχω δύο ερωτήσεις. Η μία απευθύνεται στην εκπρόσωπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και οι άλλοι στους υπόλοιπους ομιλητές. Γνωρίζουμε ότι ο αριθμός των πρόωρων θανάτων που οφείλονται στη μόλυνση του αέρα είναι πάρα πολύ ψηλή. 300.000 τέτοιου είδους θάνατοι το χρόνο. Αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι οφείλονται κυρίως από πνευμονικές ασθένειες. Προφανώς. Και φυσικά αυξάνονται σημαντικά και οι καρδιαγγειακές παθήσεις. Τι γίνεται με τους καρκίνους. Τώρα πλέον η, ε, η καρκινική όγκη είναι επιδημία Υπάρχουν εκθέσεις οι οποίες να λαμβάνουν υπόψη τις εκπομπές σαν παράγοντα καρκινογένεσης και αναφέρομαι επίσης ε, στα βενζοϊκά. Ιδιαίτερα λοιπόν τι ακριβώς γίνεται με το βενζοπυρένιο το οποίο εκπέμπεται από τη βιομηχανική κυρίως δραστηριότητα. Ένα άλλο θέμα είναι η γεωργία. Είπατε ότι η γεωργία είναι σημαντική πηγή ε, μόλυνσης. Ε, εκπλήσει σε μια πρώτη φάση γιατί η γεωργία θα έπρεπε να είναι κάτι το ε, που δεν μολύνει. Τι εκπέμπεται λοιπόν από τη γεωργία. Ε, ξέρω ότι χρησιμοποιούνται διάφορα υλικά όπως το ποτάσιο αλλά υπάρχουν και άλλοι παρά το κάλιο, αλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι ε, επηρεάζουν το περιβάλλον που εκπέμπονται από τη γεωργία. Ξέρουμε ότι αυτό έχει επηρεάσει ιδιαίτερα τον ευτροφισμό στις περιοχές που καλύπτονται από ύδατα. Στη συγκεκριμένη παρατήρηση θα ήθελα και εγώ να μιλήσω για τον ευτροφισμό. Αυτό το αντιμετωπίζουμε στα θέματα της μόλυνσης των υδάτων και μπορείτε τεχνικά να μας δώσετε κάποιες εξηγήσεις πως αυτό επηρεάζεται και επηρεάζει με τη σειρά του τη μόλυνση της ατμόσφαιρας. Θα δώσω απαντήσεις στην πρώτη ερώτηση σε σχέση με την πρόκληση ασθενειών από συγκεκριμένες αιτίες. Αναφερθήκατε στις ασθένειες στους πνεύμονες, στα καρδιαγγειακά και πρέπει να πούμε ότι στην κοινωνία μας υπάρχουν οι καρδιαγγειακές ασθένειες, αναφερόμαστε δηλαδή σε ισχυμικά επεισόδια, σε εμφράγματα, είναι φαινόμενα τα οποία κυριαρχούν στην κοινωνία μας και ακριβώς επειδή η μόλυνση στην ατμόσφαιρα συνδέεται με αυτά και η αυτοκίνηση επηρεάζει ιδιαίτερα. Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό, η βασική βλάβη ε, οι καρδιακιακές παθήσεις είναι περίπου το 80% των πρόωρων θανάτων. Ο καρκίνος ε, στους πνεύμονες είναι πολύ χαμηλότερο, 6% του συνόλου των πρόωρων μορφών θανάτου. Και αυτό γιατί υπάρχουν πολύ λιγότεροι που παθαίνουν καρκίνο στους πνεύμονες από ό,τι καρδιακιακές παθήσεις συνολικά. Και έχετε δίκιο ότι το βενζοπυρένιο είναι ένα συστατικό στο μίξ της μόλυνσης της ατμόσφαιρας το οποίο είναι υπεύθυνο για όλα αυτά. Okay, um, when it... Σχετικά τώρα με τη συνεισφορά της γεωργίας σας. Συνεισφέρει κατά 90%, 90 των εκπομπών αμμονιούχων. Αμμονίας με λίγα λόγια. Το υπόλοιπο προέρχεται από κάποιες ε, εγκαταστάσεις καύσης όπως επίσης και από την ε, ε, αυτοκίνηση. Αλλά είναι η βασική πηγή και ακριβώς η αποθήκευση και η διανομή και χρήση It's είναι κάτι το οποίο προκαλεί αυτού του είδους τις εκπομπές. Το ίδιο ισχύει και για τις εκπομπές μεθανίου, αν και δεν είμαι απόλυτα σίγουρος για το ποσοτικό κομμάτι. Πάντως συνεισφέρει και στις εκπομπές μεθανίου και συνεισφέρει επίσης κατά 5 με 10% και στις πρωτογενείς εκπομπές σωματιδίων. Και αυτό οφείλεται ίσως στην χρήση θερμαντικών σωμάτων για την αντιμετώπιση κλιματολογικών συνεπειών στα χωράφια. Τώρα η, σχέση του, ε, των αζωτούχων γενικά είναι κάτι το οποίο αλλάζει τη φύση του εδάφους και αυτό δημιουργεί προβλήματα και στον ανταγωνισμό ανάμεσα στα είδη. Κάποια είδη είναι ανταγωνιστικά σε περιοχές οι οποίες είναι φτωχές σε άζωτο και είναι το όριο αν θέλετε μερικές φορές ο δίκτυς οριακός για το ε, περιβάλλον του εδάφους όπως είναι άλλες ουσίες για άλλα επίπεδα μόλυνσης. Λοιπόν ε, κάποιες, κάποια φυτά μπορούν να ευδοκιμήσουν ενώ κάποια άλλα ε, έχουν αρνητική αντίδραση. Συνολικά όμως μειώνεται ο αριθμός των ειδών και καλύπτεται η περιοχή από, ορισμένες, από ορισμένα είδη φυτού τα οποία θεωρούνται ανταγωνιστικά στα αζωτούχα. Ε, σε περιοχές ε, ορεινές χαμηλής κάλυψης κάποια φυτά έχουν ε, αρχίσει να εξαφανίζονται, γίνονται σπάνια γιατί υπάρχει αύξηση των αζωτούχων αυτά τα φυτά είναι πιο ευαίσθητα σε επιπλέον επίπεδα αζωτούχων από ό,τι σε χαμηλότερες υψομετρικά περιοχές. Τελευταία ερώτηση για την πρώτη φάση. Yes, Ναι, ευχαριστώ. Κύριο Τέιλορ, ε, για την αστική τώρα ρήπανση, ε, μ' αρέσουν τα σχόλιά σας, αυτό που είπατε και οι απόψεις για το πόσο χρήσιμο είναι ε, να μειωθεί και η ε, απαγόρευση κινητήρων ε, πετρελαίου, δίζελ, είναι ένα από τα εργαλεία της εργαλειοθήκης. Γιατί τα ορούμενα σωματίδια είναι οι μεγαλύτεροι φωνιάδες και ευθύνονται κινητήρες του πετρελαίου, του δίζελ ουσιαστικά. Μπορώ να ξεκινήσω λέγοντας ότι ο Διεθνής Οργανισμός για την Έρευνα του Καρκίνου, που είναι της ΠΟΗ, ε, μελέτησε πάρα πολύ ε, την πετρελαιοκίνηση και έχει χαρακτηρίσει το ντίζελ καρκινογόνο για τον άνθρωπο. Ξέρουμε το μόριο σε επηρεάζει ε, την ανθρώπινη υγεία και αυτό έχει να κάνει και με το μείγμα της ατμοσφαιρικής ρήπανσης της πόλης. Βεβαίως πρέπει να ληφθεί υπόψη η πετρελαιοκίνηση. Ευχαριστώ. Θέλω και πάλι να ευχαριστήσω και τους δύο μιλητές για την πρώτη αυτή ε, ενότητα. Θα περάσουμε στη δεύτερη, το επόμενο πάνελ και θα παρακαλέσω τους τρεις επόμενους ομιλητές να έρθουν εδώ στο Προεδρείο. Σας ευχαριστώ και πάλι. Σα um, Σας ευχαριστώ. Στο δεύτερο τμήμα θα μιλήσουμε ε, για, τα ζητήματα που σχετίζονται με τη συμμόρφωση των κλάδων και έχουμε μαζί μας ε, για τις δυνατότητες μείωσης εκπομπών τον Klaus Land που είναι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Αυτοκινητοβιομηχανίας, συντονιστής των ε, εκπομπών κατά την οδήγηση σε πραγματικές συνθήκες από την Daimler στην Στουτγάρδη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που δίνετε στον κλάδο τη δυνατότητα να εξηγήσει τι έχει κάνει μέχρι στιγμής αλλά φυσικά και να εξηγήσουμε τι, θέλουμε να, τι θα θέλαμε να υποστηρίξουμε όσον αφορά και τα ζητήματα που ακούσαμε στις προηγούμενες παρουσιάσεις, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Πρώτη διαφάνεια που υπήρχε και σε μία από τις προηγούμενες παρουσιάσεις, βλέπετε τι έχει γίνει μέχρι στιγμής βλέποντας τα ευρωπαϊκά ε, πρότυπα εκπομπών για τα οξύδια του αζότου, για τη βενζίνα, για τις ε, τιμές ατμοσφαιρικών σηματίδίων. Βλέπετε τα επιβατικά οχήματα έως το επίπεδο Euro 6 και στα, αριστερά τα ΙΧ και στα δεξιά τα επαγγελματικά οχήματα. Βλέπετε ότι υπάρχουν ε, τεράστιες βελτιώσεις όσον αφορά τις εκπομπές στα νέα ε, οχήματα, στα ελαφριά τύπου, τύπου, ελαφριού τύπου και βαρέως τύπου και όπως ακούσαμε και από τις προηγούμενες παρουσιάσεις, το θέμα δεν είναι μόνο οι εκπομπές που ελέγχονται, πρέπει να εξετάσουμε και τις τις εκπομπές που πραγματοποιούνται σε πραγματικές συνθήκες. Στην πλευρά των βαρέων οχημάτων με το σύστημα μετρήσεων που ε, εφαρμόζεται αυτό που θέλω να σας δείξω είναι πώς μεταφέρουμε αυτό το φορητό σύστημα μετρήσεων από τα επαγγελματικά οχήματα στα γιοταχή. γνωρίζουν ίσως κάποιοι ότι αυτή τη στιγμή η Κομισιόν συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη και με την ε, βιομηχανία και με το, για τον κανονισμό, για την ε, οδήγηση σε πραγματικές συνθήκες για τα ελαφριά οχήματα. Γιατί χρειάζεται ένας τέτοιος κανονισμός. Ε, νομίζω ότι έγινε σαφές και στις προηγούμενες παρουσιάσεις ότι αυτό αποτελεί και τμήμα του προγράμματος για τον καθαρό αέρα και αυτό που αναφέρεται εκεί είναι ότι πρέπει να αναπτυχθεί μια νέα διαδικασία ελέγχου για να διαπιστώνονται οι εκπομπές ε, ε, οξυδίων του αζότου σε συνθήκες κανονικής οδήγησης. Είναι πλέον ε, γνωστό και έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές ότι αυτά που έχουν γίνει Βλέπετε εδώ το 2000 είχαμε το Euro 3, τον τύπο Euro 3 δηλαδή 500 μιλιγκράμμ ανά χιλιόμετρα και στο Euro 6 βλέπετε την, ε, την εξέλιξη αυτών των ε, τιμών από τα δεξιά προς τα αριστερά. Τώρα πια το πρότυπο είναι 18 μιλιγκράμμ ...80 μιλιγκράμμ Και ως βιομηχανία είναι αυτό το θέμα που μας απασχολεί και θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και συμμετέχουμε σε μια πολύ επικοδομητική και γόνιμη συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να υιοθετηθεί αυτός ο κανονισμός το συντομότερο δυνατό και για να εξελίξουμε τα, αυτοκίνητά μας ε, με βάση τις διατάξεις του. είναι, είναι, είναι το περιεχόμενο αυτού του μελλοντικού κανονισμού τώρα. Πρώτα απ' όλα, όπως εξήγησα, η πρώτη ιδέα ήταν να μεταφέρουμε αυτά τα φορητά συστήματα μέτρησης στα γεωταχή και να μετρήσουμε τα, τις εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης με αυτόν τον εξοπλισμό. Βλέπετε εδώ στα αριστερά στην εικόνα πώς το κάναμε δεν ήταν δυνατόν να, να εγκατασταθεί τέτοιος εξοπλισμός σε όλα τα αυτοκίνητα, τα Και αυτό η αυτοκινητομηχανία πίεσε ώστε να υπάρξει ένα ελαφρύ και εύκολα συνδέσιμο σύστημα ώστε να μπορούν να γίνονται μετρήσεις σε όλα τα οχήματα. Και με αυτό εννοούμε ότι κάνουμε πάρα πολλές αλλαγές, πάρα πολλές έρευνες ε, για να ε, έχουμε έτοιμα τέτοια συστήματα όταν δεθεί σε εφαρμογή αυτός ο κανονισμός. Και όταν πλέον εγκατασταθεί αυτό το σύστημα μέτρησης εκπομπών θα πρέπει να το βαθμονομήσει κανείς με δυναμόμετρο για να δει αν είναι σωστές οι τιμές. Αργότερα Βλέπετε εδώ στη δεξιά πλευρά, περνάμε από μια διαδικασία αξιολόγησης ή ένα εργαλείο ε, κανονικοποίησης και στη συνέχεια πρέπει να επιβεβαιωθούν τα πρότυπα ε, εκπομπών σε δύο τομείς, μέτρια, μέτριες εκπομπές και εκτεταμένες εκπομπές, ε, μετράμε και τη θερμοκρασία και διάφορες άλλες δυναμικές συνθήκες. Οι σημαντικοί πυλώνες αυτού του μελλοντικού κανονισμού είναι φυσικά τα όρια. Όλοι έχουμε μάλλον διαφορετική γνώμη για το τι ακριβώς συνιστά κανονική οδήγηση. Για τους μηχανικούς όμως αυτό θα πρέπει να ορίζεται σαφώς. Όχι μόνο διότι θα θέλαμε να υπάρχει μια ισότιμη εξέταση του θέματος στην Ευρώπη. Όχι είναι ευθύνη μας ο κανονισμός αυτός να ε, υιοθετηθεί και από άλλες χώρες όπως είναι η Νότια Κορέα για παράδειγμα. Γι' αυτό θα πρέπει να ε, στηρίζεται με πολύ ισχυρά στοιχεία σε μία από τις επόμενες διαφάνειες θα μπω σε κάποιες λεπτομέρειες για το πώς θέλουμε να υποστηρίξουμε την υλοποίηση αυτού του κανονισμού και εξετάζουμε το υφιστάμενο του υπάρχον σχέδιο κανονισμού, την πρόταση κοσμίου. Και στο, στην πρόταση αυτή ε, θα δείτε αν την ε, διαβάσετε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία έχει ήδη ξεπεράσει κάποια από τα στοιχεία που προβλέπονται εκεί. Στην πλευρά των ε, βαρέων οχημάτων υπάρχουν ήδη τέτοιες διατάξεις, υπάρχει ένας ε, παράγοντας ε, συμμόρφωσης 1,5 και αναμφίβολα και ο τομέας των γιοταχή θα χρησιμοποιήσει αντίστοιχα συστήματα. Αλλά συνολικά, όπως ανέφερα, το, το στοιχείο για να μπορούν να γίνουν μετρήσεις στα γεωταχή είναι αυτό το σύστημα PEMS Lite. Τα βασικά ερωτήματα για τους μηχανικούς είναι τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε κανονική οδήγηση. Για έναν μηχανικό είναι σημαντικό να γνωρίζει αν μιλάμε ε, για οδήγηση σε ανηφόρα, μιλάμε για φορτωμένο αυτοκίνητο, μιλάμε για ε, οδήγηση με φορτωμένο αυτοκίνητο σε ανηφόρα, με χαμηλές θερμοκρασίες και με τη μέγιστη επιτάχυνση. Όλα αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να διευκρινιστούν. Φυσικά όταν οριστούν αυτά τα όρια θα πρέπει να εξετάσουμε ποιος είναι ο στόχος των κανονισμών, του κανονισμού. Μπορούμε να παραπέμπουμε ή να, να ανατρέξουμε σε στατιστικά δεδομένα, αλλά εμείς ως βιομηχανία θέλουμε να πούμε ότι υποστηρίζουμε έναν φιλόδοξο κορονισμό και τον διαχωρισμό σε δύο τομείς. Τον ε, μετριοπαθή τομέα που καλύπτει το 90% της κανονικής οδήγησης αλλά και στον, στην εκτεταμένη περιοχή θα ε, υπάρχουν ε, παράγοντες CF που θα ελέγχουν την περιοχή αυτή, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα όρια, κάτι που είναι σημαντικό όχι μόνο για μας, αλλά και για όλα τα, όλες τις άλλες πλευρές που θα ελέγχουν ε, τα οχήματα, αλλά βεβαίως και για τις τρίτες χώρες. Όταν αν εξετάζουμε τα, τα λεπτομερή στοιχεία για την εκπλήρωση αυτών των διατάξεων του κανονισμού. Θα θέλαμε να σας δώσουμε ένα παράδειγμα εδώ για ένα αυτοκίνητο compact. Τι σημαίνει να πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις όπως ε, και για τα βαρέα οχήματα. Νομίζω ότι αυτό που σημαίνει είναι ότι θα πρέπει να διαμορφωθούν τα αυτοκίνητα με νέο τρόπο. Όλα αυτά που βλέπετε με κόκκινο χρώμα θα πρέπει να τροποποιηθούν, θα πρέπει να αλλάξουν γιατί ο παράγοντας ε, που ε, προβλέπεται στον κανονισμό είναι όλες αυτές οι νέες τεχνολογίες, όλοι αυτοί είναι οι εξοπλισμοί και αυτό τον λόγο θα πρέπει να αναπτύξουμε όλα αυτά τα νέα συστήματα. Φυσικά θέλουμε να το κάνουμε, αλλά όπως βλέπετε Το να γίνουν όλες αυτές αλλαγές χρειάζονται χρόνος, περίπου πέντε έτη. Σημαίνει αυτό ότι η αυτοκινητοβιομηχανία απλά θέλει να καθυστερήσει την ε, θέση σε ισχύ του κανονισμού που είναι απαραίτητο να γίνει. Όχι. Θέλουμε να εισαγάγουμε να εισαχθεί αυτός ο κανονισμός σε δύο φάσεις. Δηλαδή να ολοκληρωθεί η εφαρμογή αυτού του κανονισμού όταν θα έχουν γίνει όλες αυτές οι αλλαγές του υλικού εξοπλισμού. Τι σημαίνουν όλες αυτές οι αλλαγές. Εδώ είναι λίγο περίπλοκα τα πράγματα για να σας τα εξηγήσω. Αλλά θα προσπαθήσω να σας καθοδηγήσω στις διαφάνειες αυτές. Κατά μέσο όρο, ο κύκλος ζωής κάθε μοντέλου είναι 6 με 7 χρόνια. Στη συνέχεια, ο κλάδος λόγω και του ανταγωνισμού θα, φέρει, θα διαθέσει στην αγορά ένα νέο μοντέλο μετά από τα 6-7 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι η ανάπτυξη των οχημάτων που, εκπληρώνουν το, που πληρούν το πρότυπο Euro 6 η ανάπτυξη αυτών των οχημάτων ξεκίνησε το 2008-2009, διατίθεται αυτή τη στιγμή στην αγορά και θα ε, βγουν από την αγορά γύρω στο 2020-2021. Το να αλλάξουμε λοιπόν αυτά τα οχήματα σημαίνει ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε νέου είδους οχήματα και αυτό σημαίνει ότι το μελλοντικό μοντέλο του οποίου η ανάπτυξη έχει ήδη ξεκινήσει θα πρέπει να ξανακάνουμε όλη αυτή τη δουλειά και στο τέλος όταν λανσάρουμε ε, τις αλλαγές αυτές στα τρέχοντα μοντέλα θα σημάνουμε και το, το, το τέλος της ζωής, του κύκλου ζωής αυτών των μοντέλων. Είναι λοιπόν αδύνατον αυτή τη στιγμή να αλλάξουμε την παραγωγή και να κάνουμε τόσο σοβαρές αλλαγές από τώρα τουλάχιστον έως το 2018. Γι' αυτόν τον λόγο ε, αναφερθήκαμε ε, σε, σε αυτή την φάση, στις δύο φάσεις εφαρμογής του κανονισμού. Αυτά που, τα οχήματα που αναπτύσσουμε αυτή τη στιγμή και που πρόκειται να, βρεθ, να διατεθούν στην αγορά το 2017, αυτά μπορούμε να τα τροποποιήσουμε, να τα προσαρμόσουμε σε μια πρώτη φάση αυτού του κανονισμού RDE, γιατί πολλά από αυτά τα οχήματα ε, διαθέτουν ήδη ε, την ε, τεχνολογία ώστε να ανταποκρίνονται στις διατάξεις του κανονισμού RDE. Και με αυτό για το χρόνο εισαγωγή, όπω είπα, πρώτα απ' όλα η αυτοκινητοβιομηχανία είναι σαφή. Θέλουμε να αναπτύξουμε τα οχήματά μα με βάση τι διατάξει του κανονισμού. Αλήθεια το λέμε. Θα το κάνουμε σε δύο φάσεις όμως. Και αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει ένα ενδιάμεσο στάδιο όπου θα διατεθούν στην αγορά το Σεπτέμβριο του 2007 τα πρώτα νέα οχήματα και σε, 8, σε 5 χρόνια από σήμερα θα μπορέσουμε πλέον να λανσάρουμε αυτοκίνητα που θα ανταποκρίνονται πλήρως στις διατάξεις του κανονισμού. Σήμερα ε, εξετάζουμε την πρόταση του κανονισμού και εκεί προβλέπεται ότι το όριο το χρονικό είναι 2015 και αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος θα παραταθεί ακόμα περαιτέρω έως το 2021-2022 εμείς δεν θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε στον, στο στόχο για τον Σεπτέμβριο του 2007 Οπότε εμείς θέλουμε να έρθουμε σε διευθέτηση, με την, σε διακανονισμό με την, με την Κομισιόν για να ανταποκριθούμε και στο στόχο για τον Σεπτέμβριο του 2007. 17. Εδώ βλέπετε στα, στα δεξιά, στα πράσινα ε, κουτάκια βλέπετε ε, το βασικό σενάριο, το, στο σενάριο καθυστέρησης με το 2016 και μετά βλέπετε και τη δική μας πρόταση για την εφαρμογή σε δύο φάσεις που είναι πολύ κοντά στο σενάριο αναφοράς και βλέπετε ότι δεν υπάρχει σχεδόν καμία διαφορά μεταξύ του βασικού σενάριου και του σενάριου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ευτοκινητοβιομηχανίας. Επίσης, το 97% των σταθμών ποιότητας στη Γερμανία θα συμμορφώνονταν με τις διατάξεις του κανονισμού του 2030, αλλά θα πρέπει να αναπτυχθούν διάφορες τεχνολογίες, διάφοροι κλάδοι να κινητοποιηθούν και να δραστηριοποιηθούν ώστε να μην υπάρξουν εμπόδια στη διαδικασία. Συμπεράσματα. Η αυτοκινητοβιομηχανία ούτε καθυστερεί ούτε μπλοκάρει το RDE. Το υποστηρίζουμε. Έχουμε προτείνει ένα πακέτο, όπως το περιέγραψα, που θα ωφελήσει την ποιότητα του αέρα. Χρειαζόμαστε έναν σαφή κανονισμό όμως και είμαστε ε, πρόθυμοι να μιλήσουμε και για τα όρια που μέχρι στιγμής δεν έχουν συζητηθεί ε, αφού γίνει μια μελέτη επιπτώσεων και Όπως είπα, θα αρχίσουμε εμείς την εφαρμογή των προτάσεων μας από το 2017. Τελευταία διαφάνεια. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και εδώ βλέπετε τι είδους ωφέλη θα αποκομιστούν από το 2014, το 2017 που είναι η πρώτη φάση εφαρμογής, το πρώτο βήμα βλέπετε ότι είναι τεράστια η βελτίωση και στο τέλος θα ε, βλέπετε στο 2020 ε, την εφαρμογή συστημάτων μέτρησης εκπομπών ε, όπως υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα βαρέα οχήματα. Ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα, να περάσουμε στη Γεωργία. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Ρογκέ. Ο κύριος Ρογκέ εκπροσωπεί τα γεωργικά επιμελητήρια. Τα αγροτικά, συγγνώμη, επιμελητήρια. Daniel Roguet, agriculteur, polyculture, élevage, donc président de la Chambre d'agriculture de la Somme. Και το γεωτεχνικό επιμελητήριο. Ε, είναι η πρώτη δυνατότητα που έχω για να σας παρουσιάσω τα θέματα των, του περιβάλλοντος και της γεωργίας. Η Γεωργία εμπλέκεται σε όλα αυτά. Είναι ένα δύσκολο θέμα η σχέση μας με το περιβάλλον, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ασχολούμεθα με αυτό. Τα γεωτεχνικά επιμελητήρια είναι ένα δίκτυο. Administré par 4200 élus représentant l'ensemble des acteurs du monde agricole, rural et forestier. Λοιπόν, συμμετέχουν διάφορες κατηγορίες και για τη γεωργία και για τη δεσοκομεία. Υπάρχει η οικονομία, υπάρχει το περιβάλλον, υπάρχουν οι διοικητικοί φορείς και αυτό συνεισφέρει στον οικονομικό δυναμισμό των εδαφών. Μέχρι τώρα η γεωργία σε σχέση με το περιβάλλον ασχολήθηκε κυρίως με την ποιότητα του νερού. Έγιναν σημαντικά βήματα για να εξελιχθούν θετικά οι πρακτικές μας να λάβουμε υπόψη μας τις εξελίξεις και να χρησιμοποιήσουμε νέες πρακτικές. Σήμερα τίθεται το θέμα της ποιότητας του αέρα, της ατμόσφαιρας. Υπάρχουν τα θερμοκήπια, τα αέρια του θερμοκηπίου είναι κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα, έχει αρχίσει να δημιουργεί προβλήματα ποιοτικά και ποσοτικά. Προσπαθούμε λοιπόν να εσωτερικεύσουμε αυτόν τον παράγοντα αλλά καταλαβαίνετε ότι η γεωργία έχει και κλιματολογικές παραμέτρους, μετεωρολογικές παραμέτρους, κάτι το οποίο δημιουργεί επιμέρους διαφοροποιήσεις. Όλα αυτά έχουν και συνέπειες βέβαια και έχει σημασία να υπάρξει μια συζήτηση αλλά και μια προσπάθεια ενημέρωσης παιδαγωγικής. Έχουμε βέβαια και συγκεκριμένα όρια σε σχέση με τις παραγωγές μας σε σχέση με, την, με τον διακανονισμό της ρυθμίσης υπάρχουν πάρα πολλές οδηγίες για τα ζωτούχα, για το περιβάλλον και όλες αυτές οι ρυθμίσεις επηρεάζουν τις πρακτικές που χρησιμοποιούμε. Και σε σχέση με τα μέτρα απέναντι στις νέες οδηγίες θα πρέπει να ανταλάβουμε όλα αυτά υπόψη και να συγκρίνουμε ακριβώς τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν σε σχέση με τις δυσκολίες που υπάρχουν για να ληφθούν. Εγώ είδα ότι οι Γεωργοί μερικές φορές αντέδρασαν απέναντι σε διάφορα μέτρα τα οποία δείχνουν ότι έχουμε ένα κύκλο παραγωγής εποχιακό τον οποίο δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε σαν παράδειγμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Έχουμε επίσης και κάποια έλλειψη αναφορών, έχουμε μια έλλειψη τεχνικών πρακτικών. Έχουμε επίσης έλλειψη στον τομέα των κτηρίων. Δεν μπορούμε να βάλουμε τα ζώα μας όλα σε κτίρια. Όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη στις πρακτικές μας και θα πρέπει να τα, όπως είπα, εσωτερικεύσουμε. Έχουμε επίσης και μοχλούς σημαντικούς, τους οποίους μπορούμε να κάνουμε να δράσουν. Εξελίσσονται οι πρακτικές μας και σε σχέση με την χρήση των κτηρίων, επίσης με το χρόνο ε, βοσκής, ε, σαν παράδειγμα η κάλυψη ακριβώς κάποιων χορτολιβαδικών εκτάσεων, Sauf que toutes ces démarches-là ont un véritable coût. Je pense qu'il est important qu'on puisse avancer sur des conséquences économiques. Υπάρχουν και οικονομικές συνέπειες οι οποίες θα πρέπει να μας κάνουν να σκεφτούμε έτσι ώστε να δούμε ποια είναι τα συμφέροντα των γεωργών απέναντι σε αυτές τις πρακτικές. Το λέω ξεκάθαρα εδώ ότι η γεωργία έχει ανάγκη από ένα εισόδημα για να λειτουργήσει. Δεν μπορεί να, μην υπάρξει γεωργία χωρίς εισόδημα. Και επίσης δεν μπορούμε να μην λάβουμε υπόψη μας το περιβάλλον. Όλα αυτά λοιπόν στο παρελθόν δεν τα λάβαμε υπόψη μας, τώρα όμως πρέπει. Εγώ σαν υπεύθυνο επαγγελματίας που είμαι, θα πρέπει να προβάλλω το γενικό συμφέρον ε, στους συμπολίτες μας. Η κατάσταση του περιβάλλοντος αποτελεί μια κοινωνική κρίση και η γεωργία πρέπει να αντιλάβει υπόψη της και με συγκεκριμένο τρόπο. Αυτάρκεια τροφιμική σαν παράδειγμα είναι σημαντικό. Εμείς παράγουμε πρώτες ύλες διατροφής και ποιοτικές μάλιστα να μην ξεχνάμε ότι έχουμε επίσης ένα σημαντικό ρόλο και στον τομέα της ενέργειας, των ανανεώσιμων ε, μορφών ενέργειας, βιομάζα κτλ. Και αυτό πρέπει να γίνει με πολύ προσεκτικό τρόπο. Θα πρέπει να ανταλάβουμε υπόψη μας λοιπόν. Έγιναν προσπάθειες και όταν βλέπουμε τι κάνουν άλλες χώρες σε σχέση με τα αέρια του θερμοκηπίου κτλ. Οι πρακτικές μας έχουν αρχίσει να βελτιώνονται. Βέβαια δεν αλλάζουν όλα γρήγορα στον γεωργικό κόσμο. Έχω την αίσθηση ότι με την τεχνολογία μπορούμε όμως να δράσουμε. Αυτό είναι τμήμα και της παιδαγωγικής ενημέρωσης αλλά και της λειτουργίας της αγοράς. Οι διακυμάνσεις των τιμών σαν παράδειγμα έχουν μεγάλες συνέπειες στους γεωργούς και στην κτηνοτροφία. Ένας τομέας ιδιαίτερα ευαίσθητος, ένας τομέας που παρουσιάζει πολλούς κινδύνους. Το να υπάρξουν περαιτέρω ε, επιβαρύνσεις αυτό θα οδηγήσει σε αρνητικό, αρνητικά αποτελέσματα, αντίθετα από αυτά που αναμέναμε. Αλλά χρειάζεται ενημέρωση, χρειάζεται ευαισθητοποίηση, ακόμα και με μείωση της παραγωγής. Αυτό δημιουργεί κινδύνους και σε σχέση με τη χρήση του άνθρακα ε, και τα ε, αέρια του θερμοκήπιου. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ρεαλιστές κάποιοι στόχοι οι οποίοι δεν είναι επιτεύξιμοι και δεν είναι κατανοητοί είναι πάρα πολύ δύσκολο να επηρεάσουν θετικά τις πρακτικές μας. Πρέπει όλα αυτά να τα προσμετρήσουμε και πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας και τις οικονομικές πλευρές. Έχουμε πάρει ήδη μέτρα. Ε, ε, ενημέρωσης, κατάρτισης των γεωργών. Είμαι πεπισμένος ότι σήμερα σε σχέση με, τα, με τις συστάσεις τις οποίες πρέπει να δώσουμε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, όλα αυτά σε σχέση με τις κτηριακές μας εγκαταστάσεις, σε σχέση με τις εκμεταλλεύσεις. Ήδη ενημερώνουμε και σε επίπεδο επιμελητηρίων. Ήδη πήραμε αρκετά μέτρα στον τομέα των λοιπασμάτων. Ήδη δώσαμε συμβουλές και συστάσεις σε σχέση με, τον σωστό χρονισμό που αφορά τη μόλυνση της ατμόσφαιρας. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν στα πλαίσια μιας παιδαγωγικής διαδικασίας. Οι, οι νομικές ρυθμίσεις δεν έχουν πάντα θετικέ επιπτώσεις. Μπορεί βέβαια να ξεκαθαρίζουν ορισμένα πράγματα, αλλά στρεβλώνουν και κάποια άλλα. <clears throat> Μην ξεχνάτε ότι η γεωργία σε σχέση με το κλίμα είναι κάτι το ιδιαίτερο περίπλοκο. Αυτό αφορά και την οργάνωση της εργασίας. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Εγώ είμαι αρκετά αισιόδοξο σε σχέση με την εξέλιξη των πρακτικών μας. Αλλά είμαι πεπισμένος ότι θα πρέπει να κρατήσουμε τα επίπεδα παραγωγής μας, επίσης ε, τα επίπεδα ποιότητας της παραγωγής μας και τα περιθώρια κέρδους μας. Οι γεωργοί έχουν την τεχνολογία για να κάνουν περαιτέρω προσπάθειες, αλλά φυσικά το εισόδημά τους είναι το βασικό και απαραίτητο. Έχουμε και κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δεν γίνονται κατανοητά. Γιατί να υπάρχει μια οδηγία για το κλίμα, για τον αέρα, για τα αζωτούχα. Γιατί όχι μια οδηγία η οποία να είναι εγκάρσια, πλήρης και να είναι πιο εύκολα κατανοητή. Το είπατε άλλωστε και δεν το άκουσα αυτό ότι το 90% της μόλυνσης στην ατμόσφαιρα προέρχεται από τη γεωργία, ότι πράγματι μπορούμε να μειώσουμε αυτό το ποσοστό. Θα πρέπει όμως να είμαστε καινοτόμοι τεχνολογικά και υπολογίζω στις προσπάθειες που πρέπει να γίνουν. Σε επίπεδο λοιπόν γεωργικών επαγγελμάτων, όπως είπα, είμαστε ευαίσθητοι και θέλουμε μια εγκάρσια αντιμετώπιση και ολοκληρωμένη και όχι μια πολιτική περιβαλλοντική είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη τα χαρακτηριστικά τα ειδικά της γεωργίας και θα πρέπει να καθορίζονται ρεαλιστικά, ρεαλιστικοί στόχοι, όχι μείωση του αριθμού των ζώων. Θα πρέπει και σε ποσοτικό και σε ποιοτικό επίπεδο να είμαστε σταθεροί. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις πρακτικές μας και έτσι θα τις αλλάξουμε, κρατώντας τα εισοδήματά μας. Βέβαια το κόστος έχει σημασία. Θα πρέπει να συνοδευτούν οικονομικά οι εκμεταλλεύσεις μας για να εξυγχρονιστούν και σε επίπεδο συνθήκων ποιότητας ζωής και ποιότητας παραγωγής. Είμαι στη διάθεσή σας αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, αλλά σας λέω με κάθε ειλικρίνεια και είμαι πεπισμένος γι' αυτό ότι αντίθετα με την εικόνα μερικές φορές που έχουν οι πολίτες απέναντι στους γεωργούς, η νέα γένια ε, έχει τα τεχνολογικά μέσα και θα βοηθήσει να εξελιχθούν οι πρακτικές μας και σε οικονομικό επίπεδο και σε κοινωνικό επίπεδο. Να μην ξεχνάμε ότι είμαστε πολλές φορές ατομικής ιδιοκτησίας επιχειρήσεις με εφικτούς στόχους αλλά να μην βάζουμε στόχους που θα μας εμποδίσουν στην εξέλιξή μας. Δεν θα βοηθήσει, θα λειτουργήσει αρνητικά. Για τη συγκεκριμένη οδηγία νομίζω ότι ε, ε, λύσεις θα μπορέσουμε να βρούμε. Επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να συγκρατήσουμε το επίπεδο παραγωγής, θα πρέπει να συγκρατήσουμε τον στόχο της ε, διατροφικής ασφάλειας. Πρέπει να είμαστε επικοδομητικοί ε, και να αναζητήσουμε ο ένας ε, τις ιδέες του άλλου. Thank ευχαριστώ κύριε Ρογκέ. Τελευταίος ομιλητής για σήμερα ε, θα μας μιλήσει για ειδικά περιφερειακά θέματα και την ποιότητα του αέρα και θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Ντεμουνάρη που είναι διευθυντής, α, τώρα στα Ιταλικά, της Περιφερειακού Οργανισμού για την Πρόληψη ε, και το Περιβάλλον της Περιφέρειας Εμίλια Ρωμάν. Έβαλα τα καλύτερα Ιταλικά μου. Τα Ιταλικά σας είναι καλύτερα από τα Αγγλικά μου, οπότε θα ομιλήσω την Ιταλική, λέει ο κύριος Ντεμουνάρη. Νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή για να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε γιατί βλέπετε όταν μιλάμε για μόλυνση της ατμόσφαιρας η περιοχή της κοιλάδας του πάδου είναι μόνιμα κάτω από το κόκκινο. Έχουμε προβλήματα πάρα πολύ περίπλοκα τα οποία θα προσπαθήσω να σας δείξω έτσι ώστε να καταλάβετε καλύτερα το πώς μπορούμε να βγούμε από αυτό. Βρισκόμαστε σε μια κοιλάδα η οποία περικυκλώνεται από βουνά και δυστυχώς έχουμε πολύ μικρές, πολύ λίγες βροχοπτώσεις συνήθως και κάποιες βροχοπτώσεις οι οποίες είναι ιδιαίτερα ισχυρές σε πολύ μικρό σύντομο μάλλον χρονικό διάστημα δεν βοηθούν. Ε, έχουμε επίσης, αντιπροσωπεύουμε περίπου το 50% συνολικά του Ιταλικού ε, ΑΕΠ. Ε, Υπάρχει λοιπόν μια δραστηριότητα οικονομική η οποία δεν μας επιτρέπει στην παρούσα φάση να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις ουσίες οι οποίες μολύνουν τις περιοχές. Εμείς ε, συνεισφέρουμε κατά πολύ και σε σχέση με το οξύδιο του αζότου και σε σχέση με το όζον και σε σχέση με τα σωματίδια. Βλέπετε κάτω αριστερά πώς λόγω ακριβώς των προβλημάτων στον τομέα της βροχόπτωσης έχουμε αύξηση των σωματιδίων ε, στο, στην πεδιάδα του πάδου, ε, στην κοιλάδα καλύτερα του πάδου. Στην ουσία βλέπετε εδώ ένα τεράστιο σύννεφο από σωματίδια τα οποία εγκαθίστανται πάνω από την κοιλάδα. Όχι ότι δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα, εδώ υπάρχουν αρκετοί ε, πίνακες υπήρξε μια μείωση ε, των ε, ουσιών που μολύνουν και αναφέρομαι για την περιοχή της Εμίλια Ρωμάνια όπου σε επίπεδο θέρμανσης ε, το μεθάνιο είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιείται και σε σχέση με τις εκπομπές θείου που είχαμε προβλήματα στο παρελθόν λόγω των καυσίμων τώρα τα πράγματα έχουν διορθωθεί κατά πολύ. Έχουμε ασχοληθεί όμως λίγο με το οξύδια του αζότου, ε, τα οποία εξακολουθούν να είναι σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Βλέπετε ότι υπάρχει σε σχέση με τις εκπομπές μία μόνιμη διακύμανση και απλά στο τέλος καταλήγουμε σε έναν μέσον όρο. Τα τελευταία 15 χρόνια υπάρχει μία μείωση κατά 20%. Αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρητικά θα πρέπει να βοηθήσει την ποιότητα του αέρα, αλλά σε επίπεδο καθημερινής έκθεσης τα όρια παραμένουν υψηλά. Γιατί, για τους λόγους που είπα πριν, στην ουσία δηλαδή στο, έχουμε αρκετά μεγάλο υψόμετρο και ακριβώς ε, τα σωματίδια και οι ουσίες οι οποίες μολύνουν παραμένουν πάντα σε επαφή με την επιφάνεια του εδάφους να κάποια παραδείγματα σε κάποιες περιοχές όπως στα ε, οροπέδια της Δύσης, στην περιοχή την κεντρική και στο ανατολικό τμήμα όπως επίσης και στην ορεινή περιοχή των Απενίνων. 30 ε, μικρογραμμάρια κατά ημέρα. δεν ξεπερνάμε τις, τα ανώτατα όρια τα οποία προβλέπει η οδηγία, αλλά παρόλα αυτά ε, υπάρχουν περιοχές στις οποίες είναι μόνιμη η υπέρβαση των ορίων αυτών. Το θέμα δεν είναι μόνο για τις ε, κατοικημένες περιοχές. Οι κατοικημένες περιοχές έτσι και αλλιώς έχουν ανώτερα όρια. Έχουν υπερβεί τα όρια. Λοιπόν, αυτές αυτά είναι τα επίπεδα εκπομπών. Βλέπετε λοιπόν πως ε, οι εκπομπές ε, στα μπλε που είναι οι δικές μας από την κοιλάδα του Πάδου είναι συγκρίσιμες ε, με τις υπόλοιπες περιοχές της Ιταλίας. Στα κόκκινο βάλαμε και την περιοχή Εμίλια Ρωμάνια, η οποία και αυτή συνεισφέρει στη μόλυνση στην περιοχή της κοιλάδας του Πάδου αλλά το θέμα δεν είναι να υπολογίζουμε μόνο τις μεμονωμένες περιοχές αλλά το σύνολο της μεγάλης κοιλάδας. Λοιπόν, εδώ βλέπετε ότι αν εμείς εξετάσουμε την ποσότητα των ουσιών που μολύνουν αναπολίτη σε σχέση και με το ΑΕΠ, θα δούμε ότι φτάνουμε σε ε, ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα. Το θέμα είναι βέβαια ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πυκνότητα του πληθυσμού. Εδώ σε μία άλλη διαφάνεια βλέπει κανείς πως ε, υπάρχει και το θέμα της λεγόμενης δευτερεύουσας μόλυνσης, ε, ε, ιδιαίτερα κατά την χειμερινή περίοδο, λόγω ακριβώς της καύσης για θέρμανση. Υπάρχουν και άλλα δευτερεύοντα συστατικά από οργανικά αεροσόλ, τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά αν δείτε ότι και σε περιοχές όχι μόνο αστικές αλλά και σε περιοχές γεωργικές είναι ιδιαίτερα υψηλές αυτές οι μορφές μόλυνσης. Εδώ βλέπετε τις αιτίες, τις πηγές αυτών των μορφών της ε, μόλυνσης για την Εμίλια Ρωμάνια, την περιφέρεια. Η πρώτη αιτία αν θέλετε προέρχεται από τις μεταφορές και από την θέρμανση των αστικών περιοχών. Αν δούμε για τα οξύδια του αζότου βλέπουμε ότι το 75% προέρχεται από τις μεταφορές και τα υπόλοιπα προέρχονται από την παραγωγή ενέργειας και από τις βιομηχανικές δραστηριότητες. Βλέπει κανείς εδώ ότι οι πιο σημαντικές πηγές πάνω στις οποίες θα πρέπει να εργαστούμε είναι η αυτοκίνηση και η θέρμανση και σε ορισμένες περιοχές η βιομηχανία. Αλλά δεν είναι η βιομηχανία η περίπτωση στην οποία μπορούμε να παρέμβουμε με αποτελέσματα. Έχουμε ακριβώς κάνει προσπάθειες για την εξυγίανση του αέρα της περιοχής αυτής, κάποιες προτάσεις, βλέπετε τις μικρές ε, ε, περιοχές με κόκκινο, όπου σε μόνιμη βάση ημερήσια υπάρχει μια ε, μόνιμη υπέρβαση των ανωτάτων ορίων, με κίτρινο χρώμα είναι οι πιθανές υπερβάσεις και ε, με πράσινο εκεί όπου είναι σπάνιες οι υπερβάσεις. Το καλύτερο στο οποίο μπορούμε να καταλήξουμε είναι ε, ο κάτω δεξιά πίνακας, πράσινος και κίτρινος. Βλέπουμε εδώ ότι δεν έχουμε μία ενιαία περιοχή αλλά έχουμε διαφοροποιήσεις και υπάρχουν ε, δυστυχώς δυνατότητες και για χειροτέρευση σε ορισμένες περιοχές. Έχουμε δημιουργήσει μέσα τα οποία μας επιτρέπουν να κάνουμε αναλύσεις κόστους-οφέλους για να δούμε ποιες είναι οι πρακτικές που θα μας βοηθήσουν να εκμεταλλευτούμε σωστά τα εδάφη μας, χωρίς συνέπειες για το περιβάλλον. αν χρησιμοποιήσουμε περιορισμένα οικονομικά μέσα, αν χρησιμοποιήσουμε μόνο το 20% των διαθεσίμων, μπορούμε να περάσουμε σε σημαντικές μειώσεις, εκτός από ορισμένε περιοχές γύρω από την πόλη της Πιασέντζα, όπου οι αξίες, οι δείκτες παραμένουν ιδιαίτερως υψηλοί. Η περιοχή λοιπόν αυτή προσπαθεί να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα συνολικότερο, για να το κάνει αυτό έχει συνδυάσει μια ολόκληρη σειρά δημοσίων υπηρεσιών και δημοτικών υπηρεσιών. Πρέπει να μιλήσουμε ε, ε, για τη μείωση των θιούχων κατά 47% και των αζωτούχων κατά 36%. Δηλαδή ο στόχος είναι πάρα πολύ ψηλός. Παρ' όλα αυτά έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες τα τελευταία 10 χρόνια με τα διάφορα τοπικά προγράμματα στα οποία αναφέρθηκα πριν συμμετέχουν όλοι οι δήμοι και οι κοινότητες της περιφέρειας σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο έχει χρειαστεί και σημαντικά ύψη χρηματοδότησης. Παρ' όλα αυτά παραμένει ένα πρόβλημα ότι έχουμε να κάνουμε με μια περιοχή η οποία αφεαυτής από μόνη της η περιοχή αυτή δεν μπορεί να καταφέρει να περάσει στα αποτελέσματα τα επιθυμητά γιατί η μόλυνση των περιφερειών και των γειτονικών είναι κάτι το οποίο ανταλλάσσεται ανάμεσα στις περιοχές. Η μία επηρεάζει την άλλη. Ε, και δώσατε το παράδειγμα για την Ολλανδία. Ε, και στην περιοχή της κοιλάδας του Πάδου η ανταλλαγή αν θέλετε προβλημάτων μόλυνσης είναι δεδομένη με τις όμορες περιοχές. Είναι ένας από τους λόγους λοιπόν για τους οποίους οι περιφέρειες δεν έχουν αυτόνομα και πάρα πολλά, πολλά περιθώρια γιατί γνωρίζετε ότι από την κοιλάδα του Πάδου περνούν και όλοι οι αυτοκινητόδρομοι που συνδέουν τον νότο με το βορρά της Ευρώπης με ό,τι αυτό συνεπάζεται, συνεπάγεται σε επίπεδο κυκλοφορίας. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν για την περιφέρεια να επηρεάσει ε, πάνω από ένα ποσοστό τουλάχιστον ε, την ε, διαδικασία μείωσης της μόλυνσης. Είπαμε ότι η αυτοκίνηση είναι βασικό πρόβλημα. Λίγα πράγματα. Εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί αν δεν δούμε συνολικά τις δράσεις τις οποίες πρέπει να αναλάβουμε σε πολιτικό επίπεδο θα αντιμετωπίσουμε περαιτέρω προβλήματα. Στην Ιταλία χρηματοδοτήθηκε η ε, ανακαίνιση αν θέλετε και ο εξυγχρονισμός ε, του συνόλου των αυτοκινήτων, ιδιαίτερα επαγγελματικών. Αυτό είναι σωστό. Ταυτόχρονα χρηματοδοτήσαμε την αντικατάσταση ενός παλαιού τύπου ε, στόλου αυτοκινήτων με νέα αυτοκίνητα αλλά πετρελαιοκίνησης αυτή τη φορά. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχουμε ουσιαστικά μια πολύ μικρότερη βελτίωση από την αναμενόμενη. Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα της βιομάζας και της παραγωγής βιομάζας, της μεσοκαύσης. Είναι μια καλή πρακτική, είναι σωστή πρακτική σε επίπεδο διαχείρισης γεωργικής και παραγωγής διοξιδίου του άνθρακα, αλλά για την ποιότητα του αέρα είναι καταστροφικό γιατί βάζουμε έτσι στην ατμόσφαιρα τεράστιες ποσότητες μικροσωματιδίων. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες και βλέπετε ότι από την καύση γενικότερα στην Λομβαρδία υπάρχει παραγωγή βενζο ε, πυρενίου ιδιαίτερα υψηλή. Un determinato impianto di abbattimento che ci consente di ridurre le emissioni o se le mettiamo αυτό είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί ε, πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν μικρά θερμαντικά σώματα με λειτουργούν με ξύλο και τα οποία έχουν χειροτερεύσει την κατάσταση γιατί αυξάνεται η χρήση τους. Ένα θετικό στοιχείο ε, στο οποίο έχουμε σταθεί τα τελευταία χρόνια στην Ιταλία αλλά για το οποίο ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι δράσεις στον τομέα της ποιότητας του αέρα είναι το θέμα της θέρμανσης των κτηρίων. Υπάρχουν περιοχές στο Τρεντίνο, στον, Άλτο Άντιτζε που έχουν δώσει την δυνατότητα να χρησιμοποιούμε ε, καυστήρες 10 φορές πιο αποδοτικούς <coughs> και σε περιοχές ακόμα πιο ψυχρές από την Εμίλια Ρωμάνια. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να κάνουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό των εκπομπών ε, στην κοιλάδα του πάδου. Επιτρέπει να πετύχουμε αποτελέσματα τα οποία είναι επιθυμητά, να μειώσουμε την, τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε, και είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει και τους πολίτες ε, να κάνουν ε, εξοικονομήσεις χρημάτων γιατί καταναλώνουν ε, λιγότερα χρήματα εφόσον χρειάζονται λιγότερο καύσιμο. Τελικά, αυτό το οποίο θα ήθελα να ληφθεί υπόψη είναι ότι εμείς στην κοιλάδα του Πάδου έχουμε εκπομπές αντίστοιχες με την υπόλοιπη Ευρώπη και με τις εκπομπές της Ιταλίας είμαστε περίπου στο μέσον όρο. Όταν μιλάμε για εκπομπές της κοιλάδας του Πάδου εννοούμε περίπου τις εθνικές ε, εκπομπές. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να βρούμε ένα καλύτερο τρόπο όλες αυτές τις δράσεις να τις ολοκληρώσουμε και να τις συνδυάσουμε σωστά. Αυτό το οποίο θα ήθελα επίσης να πω όταν βλέπουμε αυτά τα κόκκινα σημεία ε, δεν πρέπει να απογοητευόμαστε και να λέμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Προσπαθούμε και σε σχέση με το πρόγραμμα LIFE να, να βάλουμε σε εξέλιξη συγκεκριμένα προγράμματα. Ακολουθούμε πολιτικές στην κοιλάδα του Πάδου έτσι ώστε να βελτιώσουμε την κατάσταση μέσω της χρήσης των προγραμμάτων βελτίωσης ε, της ατμόσφαιρας. Δεν μπορούμε να είμαστε αδρανείς αυτό είναι ε, σαν συνέπεια είχε όλες οι τοπικές αρχές να συνεργάζονται έτσι ώστε να βελτιώσουμε και τα, στους δείκτες και τις πολιτικές μας και να αντιμετωπίσουμε συνολικά, σφαιρικά την περιοχή του πάδου και όχι σαν ένα σύνολο επιμέρους μικρότερων περιοχών δύσκολα συνεργάσιμων. Ευχαριστώ. very Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και εδώ ολοκληρώνονται οι παρουσιάσεις του δευτέρου πάνελ. Έχουμε ένα τέταρτο περίπου για ερωτήσεις. Ε, τα μέλη, η κυρία Κονέσσα. Ε, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Ντεμουνάρη για την τελευταία παρουσίαση, διότι και εγώ κατάγομαι από την Μοραβία Σιλεσία στην Τσεχική Δημοκρατία που είναι η πιο μολυσμένη περιοχή. Ε, και επί σειρά ετών ε, η βιομηχανία ρήπανε ε, αλλά όχι ε, κατά κύριο λόγο ε, οι μεταφορές ήταν εκείνες που ρίπαιναν περισσότερο από τη βιομηχανία γιατί δεν μπορούσαμε να βγάλουμε την κίνηση από τις πόλεις. Ε, και χάρηκα που σας άκουσα ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και σε άλλες χώρες δηλαδή, όχι μόνο στη δική μου. Θα ήταν χρήσιμο να επικεντρωθούμε σε μια ανταλλαγή πληροφοριών για να δούμε ποιες είναι οι βέλτιστες τεχνολογίες, ιδιαίτερα για μικρές εγκαταστάσεις καύσης ε, στα νοικοκυριά που είναι σόμπες βασικά και καυστήρες ε, για να δούμε πώς θα ξεφύγουμε. Όταν μιλάμε για σωματίδια 2,5 ή ε, σωματίδια PM10 έχει σημασία να πούμε ότι είναι αντίστοιχα τα προβλήματα και τα ίδια. Και να ανταλλάξουμε λοιπόν πληροφορίες και πρακτικές σε πιο τακτή βάση έχει σημασία να μην επανεφευρίσκει ο καθένας τον τροχό, αλλά να διδαχθούμε από τη δική σας εμπειρία. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε για τις μεταφορές. και για τις νέες δοκιμές ε, και τους νέους κινητήρες. Ε, τώρα μιλώ στον εκπρόσωπο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Γιατί δεν επικεντρωνόμαστε περισσότερο ακριβώ σε εναλλακτικέ πηγές καυσίμων για παράδειγμα, ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα ε, με υδρογόνου ας πούμε, υγραερίου, βιολογικό αερίου. Όλα αυτά είναι εναλλακτικά καύσιμα που κατά την άποψή μου είναι ελπιδοφόρα και μια νέα προοπτική για το μέλλον, για να βγούμε σταδιακά, να ξεφύγουμε από τον ντίζελ και την πετρελαιοκίνηση. Τουλάχιστον στην Τσεχική Δημοκρατία Καμιά φορά δεν έχουμε αρκετές δυνατότητες ε, να διευρύνουμε τη χρήση αυτών των οχημάτων. Είναι περιορισμένη η εμβέλεια. Έχει να κάνει και με τις συνήθειες των καταναλωτών. Πώς βλέπετε το μέλλον εσείς για εναλλακτικά καύσιμα και εναλλακτική κίνηση των αυτοκινήτων, γιατί νομίζω αυτή είναι η προοπτική για το μέλλον. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα ομαδοποιήσω τις ερωτήσεις ε, πριν δώσουμε το λόγο για τις απαντήσεις. Ο κύριος ε, Μπραν, θα ήθελα να ρωτήσω ε, τι πιστεύετε για το ρόλο των δασών και για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, αλλά και για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να αυξήσουμε τη δασική κάλυψη στην Ευρώπη και αν ναι, Ποια είναι τα υπέρ και ποια τα κατά αυτής της περίπτωσης. Ευχαριστώ. Κάθριν, uh, Thank you, my... Ε, ζητώ συγγνώμη γιατί θα φύγω σε λίγο. Ε, κύριε Πέρντε, θέλω να ρωτήσω για τη Γεωργία κάτι. Γιατί θα πρέπει να έχουμε ρεαλιστική νομοθεσία, ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη. Το κατανοούμε όλοι και πόσο σημαντική είναι η Γεωργία για την ευρωπαϊκή οικονομία. Έχουμε επίγνωση αυτού και πρέπει. Όμως, δεν έχω καταλάβει πάρα πολύ καλά. Μπορείτε να μας πείτε ποια στοιχεία της νομοθεσίας είναι τελείως ανεδαφικά ποια είναι τα ρελιστικά μέτρα που σχεδιάζει ο γεωργικός τομέας για να μειώσει την παραγωγή μεθανίου και αμμονίας. Γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα και αναγκαιότητα μάλιστα να βάλετε κι εσείς ε, το λιθαράκι σας. Τι θεωρείτε λοιπόν απολύτως ανέφικτο και τι εφικτό. Να σας δώσουμε το λόγο πρώτα να απαντήσετε εσείς κύριε Λάγκε. Yes, thank you very much. Um, not... Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αν κοιτάξετε το στόχο για το 2020, για το στόλο, αυτός μπορεί να επιτευχθεί μόνο με νέες τεχνολογίες όπως τα ευρυδικά, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κτλ. Οπότε, επαναρχόμενο στο ερώτημά σας, ναι, ο κλάδος γνωρίζει ότι όλες αυτές οι τεχνολογίες θα πρέπει να διατεθούν στους καταναλωτές, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να αποφασίσουν ποια είναι η καλύτερη για τον καθένα επιλογή, για τη δική του, για, ο καθένας ξεχωριστά, για την καθημερινή του οδήγηση. Ωραία. Για τα δάση. Ίσως μπορείτε, κύριε Ρογκέ, να μας μιλήσετε. <laughs> Euh, ε, τώρα ε, βέβαια ε, το θέμα αυτό είναι επίκαιρο για τα δάση, αλλά να σας πω πρώτα για τη γεωργία. Θέλουμε να έχουμε μία ε, ισορροπία ανάμεσα στην παραγωγή τη γεωργική και τη δασοπονία. Γιατί καταλαμβάνει γεωργικές γέες η δασοπονία και έχει, το ρόλο της να παίξει. Ε, αλλά δεν ξέρω αν θα πρέπει να επεκταθεί αυτό. Ε, γιατί ε, αλλάζουν χρήση οι γέες και δεν είναι διαθέσιμες για τη γεωργία. Αλλά θα πρέπει να συνυπολογίζεται στη λύση του προβλήματος του διοξιδίου του άνθρακα. Ευχαριστώ. Σε σχέση με αυτό που είπε η κυρία Μπίρντερ, πού θεωρείτε ότι βλάπτει η πρόταση τη Γεωργία και δεν είναι ρεαλιστική. Πιστεύω ότι στην πράξη εμείς δεν θέλουμε να μας επιβάλλουν πράγματα ανέφικτα για τη ε, μείωση της αμμονίας. Είναι πάρα πολύ υψηλή η στόχη και ε, ε, σε σχέση με τις πρακτικές τις δικές μας τις περιοριζόμαστε. Δηλαδή πρέπει να έχουμε κάπου ε, λιπάσματα για την παραγωγή μας, εφόδια για τη γεωργία, για να μπορούν οι, εργάτες, οι αγρότες συγγνώμη, να καλλιεργούν. Δεν μπορούμε να έχουμε στόχους μείωση 30, 40 και 50% μέχρι το 2020, το 2050 και χρειάζεται κάποια αλλαγή και ε, κάποια ε, σταδιακή ε, προσαρμογή και να μειωθεί το κόστος της πρακτικής αυτής. Να υιοθετήσουμε νέες τεχνολογίες. Εγώ είμαι υπέρ της έρευνας για νέες ποικιλίε, για νέα παραγωγή, για να μειωθούν τα εφόδια και τα λοιπάσματα, αλλά να αλλάξουν και οι πρακτικές για πολύ συγκεκριμένα θέματα. Παράδειγμα, έχουμε συγκεκριμένες πρακτικές καλλιέργειες ανάλογα με τις εποχές του χρόνου. Έχει βγει μια απόφαση για περιορισμό των λιπασμάτων την άνοιξη. Θυμίζω ότι οι καλλιέργειές μας έχουν ειδικέ ανάγκες σε ειδικέ εποχές. Βέβαια μπορούν να αλλάξουν οι πρακτικές ε, για ε, να μην ε, γίνονται ας πούμε ψεκασμοί το πρωί, αλλά δεν μπορείς να πεις όλη την άνοιξη δεν θα χρησιμοποιώ λίπασμα. Ή ότι έχει να κάνει ακριβώς με τους ψεκασμούς ε, που σήμερα είναι πάρα πολύ ε, ρυθμισμένη. Αν θέλουμε τώρα να ε, βάλουμε ένα πολύ στενό κορσέ, αυτό θα σημαίνει ότι αυτόματα αυξάνεται η επένδυση διότι αυξάνεται το κόστος αποθήκευσης. Ήδη έχουμε κάποιες πρακτικές για να ε, χρησιμοποιούμε ε, πολύ γρήγορα την ε, κοπριά στα χωράφια και να μην την αποθηκεύουμε. Το 2013 μας χορήγησαν μια ειδική εξαίρεση γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα αποθήκευσης σε τάφρους και σιλό. Δεν έχουμε επίσης πραγματικά στοιχεία αναφοράς για να βασιστούμε σε αυτά και να αλλάξουν κάπως τα κριτήρια. Ευχαριστώ. Η κυρία Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις στον καθηγητή Ντεμουνάρη. Και εγώ προέρχομαι από την κοιλάδα του Πάδου, στην περιοχή με την οποία ασχοληθήκατε και γνωρίζουμε όλα αυτά τα δεδομένα περίπλοκα και δύσκολα Ίσως ε, να μου δώσετε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες. Και, ε, Αναφερθήκατε ότι όχι μόνο οι αστικές περιοχές έχουν πρόβλημα. Για να καταλάβω καλύτερα, γιατί υπάρχουν αυτές οι συγκεντρώσεις ιδιαίτερα υψηλές σε σχέση με τις άλλες περιοχές ε, της κοιλάδας και αν η αυτοκίνηση είναι πρόβλημα όχι μόνο στις αστικές περιοχές βέβαια, αλλά συνολικότερα και σε σχέση με την προσπάθεια την οποία κάνουμε. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν περιοχές όχι μόνο στην Ιταλία που αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσκολίες και όπως η περιοχή του Πάδου αντιμετωπίζουν μειονεκτήματα σε σχέση με άλλες περιοχές. Υπάρχουν κάποια τεχνικά στοιχεία τα οποία να μας επιτρέψουν να διαφοροποιήσουμε λίγο τη δράση μας απέναντι σε αυτές τις περιοχές που δεν θα πρέπει φυσικά όλες να αντιμετωπίζονται οι ίδιες. Δεν έχουμε να κάνουμε μια ορεινή γαλλική περιοχή στην οποία υπάρχει πολύ μεγαλύτερη διασπορά των πηγών μόλυνσης. Είναι αλήθεια ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν είναι όλες περιοχές τις ίδιες και σε επίπεδο φύσης των ουσιών που μολύνουν, οι οποίες παραμένουν πολύ περισσότερο στο εσωτερικό της κοιλάδας ε, τα, μέτρα, ε, τα, τα στοιχεία καταμέτρησης δείχνουν ότι όταν υπάρχουν ε, οξυμένες κλιματολογικές περιοχές τα πράγματα εξελίσσονται με διαφορετικό τρόπο αν βρίσκεται κανείς στο βάθος της κοιλάδας σε ενδιάμεσο έδαφος ή σε υψηλό. σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούμε να ασχοληθούμε με προβλήματα αποτελεσματικά πρωτογενούς μόλυνσης, ενώ τώρα έχουμε δευτερογενούς μόλυνσης όπως τα οξύδια του αζότου και οι άλλες πτυτικές ουσίες. Είναι προϊόντα καύσης ουσιαστικά και σε αυτή την περίπτωση όταν βρίσκονται στην ατμόσφαιρα αντιδρούν και δημιουργούν την μόλυνση σε δευτερογενές επίπεδο. Γι' αυτό ακριβώς η περιφέρεια από μόνη της κάνει αυτό το οποίο μπορεί. Αλλά νομίζω ότι όλα τα προβλήματα της περιοχής ε, δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ένα πείραμα που λέει θα κλείσουμε όλους τους διακόπτες και θα δούμε τι θα γίνουμε. Αν πραγματικά δεν γινόταν τίποτα στην περιοχή μας και αν δεν ήταν ένα μεγάλο δάσος και αν δεν κατοικούσε κανείς τότε στην ε, Πιατσέντσα σαν παράδειγμα ίσως να φτάσουμε στα επίπεδα τα οποία προβλέπουν τα κοινοτικά μέτρα. Έχει σημασία λοιπόν να δούμε και τις ε, συνέπειες των γειτονικών πηγών μόλυνσης και η αυτοκίνηση τώρα είναι δυστυχώς ε, μια βασική πηγή μόλυνσης, διαπερνά την περιοχή μας ίσως λίγο χονδρικά να το πω, το 1 τρίτο προέρχεται από τους αυτοκινητοδρόμους, 1 τρίτο από τις πόλεις και 1 τρίτο από τους περιφερειακούς δρόμους. Δηλαδή, όταν εσείς προσπαθείτε να αποκλείσετε τα αυτοκίνητα από την πόλη, όταν παίρνετε άλλα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας, και προσπαθείτε να διευρύνετε τις περιοχές ελεγχόμενης κυκλοφορίας, στην ουσία ελέγχετε τις εκπομπές ε, ε, πρωτογενούς φύσεως εσωτερικό των πόλεων. Αλλά αυτό δεν μας λύνει το πρόβλημα που έχουμε εμείς γιατί δεν ασχολείστε παρά μόνο με το 1 τρίτο των πηγών μόλυνσης. Και αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και γι' αυτό οι περιφέρειες θα πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους και πέρα από τις περιφέρειες θα πρέπει να υπάρξει επιτέλους ένα Ιταλικό κράτος το οποίο να προσπαθήσει να διαχειριστεί καλύτερα την διακίνηση κυρίως των εμπορευμάτων με λιγότερες βλάβες για την κοιλάδα του Πάδο. Τώρα. Τώρα σε επίπεδο συστάσεων ή συμβουλών ε, εξαρτάται. Εμείς έχουμε καταλήψει τις εμπορικές μεταφορές, τις υδρομικές. Τις έχουμε μεταφέρει όλες τις οδικές μεταφορές. Έχουμε κάνει τεράστια κέντρα διαμετακομιστικά, αποκλειστικά για φορτηγά μεταφορικά. Και έχουμε εγκαταλείψει με λίγα λόγια το τρένο, τον σιδηρόδρομο και σε επίπεδο επίσης κατοικιών μπορούμε να κάνουμε τεράστιες προσπάθειες για να καλύψουμε κάποιες, ε, κάποια κενά τα οποία περιοχές όπως τον Τρεντίνο έχουν ήδη σε ένα μεγάλο βαθμό κλείσει. Ε, τώρα ε, στη Ραβένα τώρα υπάρχουν κάποια επιπλέον προβλήματα γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πετροχημικό δηληστήριο Υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένα θέματα σε συγκεκριμένες περιοχές. Το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να δούμε την περιφέρεια σαν μακροπεριφέρεια. Ευχαριστώ. Και με αυτό τέλειωσε ο χρόνος μας. Οπότε ως εισηγήτρια θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους τους προσκεκλισμένους μας τους ευρωβουλευτές που υπέβαλαν ερωτήσεις και όλους τους υπόλοιπους που παρευρέθησαν εδώ για την υπομονή σας. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα που το γνωρίζετε και οι εργασίες μας θα καταλήξουν ε, σε παρουσίαση έκθεση στην Επιτροπή στις αρχές του επόμενου ε, έτους. Είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ περίπλοκο ζήτημα, αλλά είναι και πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά την ε, υγεία και το περιβάλλον. Οπότε προσβλέπω στη συνεργασία σας στους επόμενους μήνες. Σας ευχαριστώ και πάλι όλους που ήσασταν εδώ και σας εύχομαι καλή επιστροφή στα σπίτια σας.